Chers collègues, je vous demande de prendre place, que nous puissions. Euh, Καθίστε συνάδελφοι, για να ξεκινήσουμε μα. Et je suis heureuse. Είμαι πολύ ευτυχή που έχουμε μεταξύ μα μετα, μετά από την συνάντηση που είχαμε στην ε, Μαδρίτη, για όσου τουλάχιστον ήταν, ε, συμμετείχαν στην ε, αντιπροσωπεία που είχαμε, και συναντήσαμε λοιπόν την Ισπανική Προεδρία ε, με πολύ ειδικό τρόπο. Γιατί, τι να σας πω, είναι η πρώτη Προεδρία η οποία στην ουσία ζει ε, με όρους εφαρμογής συνθήκης της Λισαβόνας και όσον αφορά τα θεσμικά και όσον αφορά τα νομικά ζητήματα. Θέση σε ισχύ κυρίως της ρήτρας που μας ενδιαφέρει, της λεγόμενης οριζόντιας ρήτρας. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν είμαι πολύ ευτυχής που εξ ονόματος των συναδέλφων ε, σας υποδέχομαι σήμερα το πρωί εδώ. Η Ισπανική Προεδρία επίσης ε, πρέπει να αντιμετωπίσει μια ειδική κατάσταση η οποία όσον αφορά τα θέματα το που μας ε, προβληματίζουν εδώ είναι δυστυχώς απολύτως επίκαιρα. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερη κρίση και κρίση που στην Ισπανία παίρνει απολύτως ιδιαίτερες διαστάσεις. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σας προτείνω να πάρετε ε, τον λόγο ο ένας μετά τον άλλον ε, με την σειρά με την οποία είστε καθισμένοι. Και θα ακολουθήσει μετά από τις τρεις παρεμβάσεις σας ε, μια γενική συζήτηση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Θελεστίνο Κορμπάτσο, Υπουργό απασχόληση και Μετανάστευσης και θα σας δώσω τον λόγο για 15 λεπτά. Ε, στον κύριο Υπουργό, λοιπόν, απασχόληση και Μετανάστευσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και θερμά ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, Καλημέρα και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την παρουσία μου εδώ στην Επιτροπή σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητε τη Ισπανική Προεδρία σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων και προστασία. Η πρόσφατη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία για ένα μεγαλύτερο άνοιγμα αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη και μια Ευρώπη πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Η Ισπανική Προεδρία κατά το πρώτο αυτό εξάμεινο του 2010 θα εκτυλιχθεί σε ένα σενάριο με πολύ σημαντικά γεγονότα. Καταρχήν ε, θα έχουμε τις συνέπειες από τη θέση ισχύ της νέας συνθήκης της Λισαβόνας και θα έχουμε και νέα θεσμικά όργανα που σίγουρα θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα νέο Συμβούλιο και μια ανανεωμένη, αναζωογονημένη εξωτερική πολιτική. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ε, προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, ενισχύθηκε με ένα σημαντικό εργαλείο, αυτό της συναπόφασης, που αυξάνει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Κάτι που μετατρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα συνομοθέτη στους περισσότερους τομείς των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2010 διεκπεραιώνεται και η στρατηγική της Λισαβόνας που εγκρίθηκε το 2000. Η στρατηγική αυτή ήταν εμπλουτισμένη με φιλόδοξους στόχους που παρόλο που δεν υλοποιήθηκαν στο έπακρο θα πρέπει να την αξιολογήσουμε για τη συμβολή της στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που διανύουμε δυστυχώς παρεμπόδισε την πλήρη υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή, όμως, Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να αντιδράσει για να αποφύγει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάρρευση. Παρ' όλα αυτά η κρίση επηρέασε όλους τους οικονομικούς κλάδους και προκάλεσε μια σημαντική απώλεια παραγωγικού ιστού, κάτι που οδήγησε στην κατάργηση εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Ε, επλήγησαν ιδιαίτερα οι νέοι με τον κίνδυνο να ματαιωθούν οι προσδοκίες μιας ολόκληρης γενιάς. Η έξοδος από την παρούσα κρίση σε ένα πλαίσιο σημαντικών και βαρισίμαντων μάλλον θεσμικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις για την Ισπανική Προεδρία και τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Προεδρία θα συμβάλλει για να ε, δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, ε, να αναζωογονηθεί η οικονομία και να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία. Άλλωστε αυτή είναι η κοινή στόχη του τρίου, των τριών προεδριών, Ισπανίας, Βελγίου και Ουγγαρίας. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης θα πρέπει πρώτα απ' όλα να χαράξουμε και να κατασκευάσουμε ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει μια συντονισμένη πολιτική όθηση. Και το εργαλείο αυτό θα είναι σίγουρα η στρατηγική του 2020. Μια στρατηγική που θα πρέπει να αυξήσει την, ανταγωνιστικότητα και να ενισχύσει την οικονομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα είναι πιο αηφόρο και θα στηρίζεται στην κατάρτιση και στη γνώση θα δημιουργεί δε θέσει απασχόληση και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Του τελευταίου μήνε το χρηματοπιστωτικό σύστημα άρχισε να ανανύπτει και βελτιώθηκε η ρευστότητα των πιστώσεων. Παρόλο που οι μακροοικονομικοί δείκτες έχουν μια θετική ανάπτυξη, δυστυχώς εξακολουθούν να χάνονται θέσεις απασχόλησης. Οπότε η στρατηγική του 2020 θα πρέπει να δώσει δύο ίδια απαντήσεων. Μία βραχυπρόθεσμη, που στόχο θα έχει τη βελτίωση της κατάστασης στην απασχόληση και μία μέσο και μάκρο πρόθεσμη που θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο ισχυροί και πιο ανταγωνιστικοί σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις αυτές, χρειαζόμαστε δύο στοιχεία που έχουν αποφασιστική σημασία κατά τη γνώμη μας. Θα πρέπει καταρχήν να διατηρήσουμε τα εθνικά σχέδια εναυσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναζωογονήσουμε την οικονομία και να διατηρήσουμε τι θέσει απασχόληση. Δεύτερον, θα πρέπει με αποφασιστικό τρόπο και πυγμή να προωθήσουμε το συντονισμό μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και του ε, κοινωνικού εταίρου, προκειμένου ε, να καταστεί προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων απασχόληση. Η στρατηγική θα πρέπει να βρει σύμφωνο στους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών και φυσικά να στηριχθεί στη συνεργασία των θεσμικών οργάνων. Ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει για να κατασκευάσουμε από κοινού τα θεμέλια της μελλοντικής στρατηγικής για το 2020. Μια στρατηγική που θα διατηρήσει και θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης μέσω κάποιων δραστηριοτήτων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την κατάρτιση και τα προσόντα των εργαζομένων. Θα προωθήσει αγορές εργασίας που θα δίνουν ενάψματα στην προσφορά εργασίας, θα προωθεί νέες πηγές απασχόλησης, κυρίως ε, αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη φροντίδα των ανθρώπων ή τις νέες τεχνολογίες της ε, πληροφορίας και επικοινωνίας. Επίσης, θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία επιχειρήσεων, ε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της απασχόλησης, ενισχύοντας κάποιες ενεργές πολιτικές. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην κοινωνική οικονομία και να πατάξουμε την ε, παραοικονομία και την ε, λαθρεργασία. Τα εργατικά μοντέλα θα πρέπει να στηρίζονται στις αρχές του flex security, ευελιξία και ασφάλεια, προκειμένου να δώσουμε μια κατάλληλη λύση στις ιδιαιτερότητες των εθνικών οικονομιών. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις στην καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης αποτρέποντας τη μακροχρόνια ανεργία. Έτσι, θα εστιάσουμε τις πολιτικές μας προς τα, τις ομάδες του πληθυσμού που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Και οι νέοι ε, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρός. Θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιους μηχανισμούς ευελιξίας που θα δίνουν έμφαση όμως και στο θέμα της ασφάλειας ξεκινούμε μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί, όχι μόνο στη χάραξη της νέας στρατηγικής του 2020, αλλά και στην εφαρμογή των ε, στόχων που θα συμφωνήσουμε. Οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνδρες και γυναίκες, σε μια τέτοια οικονομική κρίση δεν περιμένουν από την στρατηγική μια απλή διακήρυξη αξιών χωρίς απτές δεσμεύσεις για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν. Και αυτή ήταν μία από τις αδυναμίες της στρατηγικής της Λισαβόνας, ότι απομακρύθηκε από τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό στη νέα φάση που διανύουμε της ε, στρατηγική για το 2020 θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση και τον κοινωνικό διάλογο, ε, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης που θα, γίνει, θα ξεκινήσει αύριο στη Βαρκελόνη όπου θα εκπροσωπείτε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Προέδρου σας. Εκεί θα γίνει μια συζήτηση που σίγουρα θα συνεχιστεί στην άτυπη διάσκεψη κορυφής του Φεβρουαρίου και στο έψικο του Μαρτίου, καθώς και στο Εαρινό Συμβούλιο. Στη διαδικασία αυτή όλοι οφείλουμε και δυνάμεθα να συμβάλλουμε. Για να υπεργούμε αυτή την παγκόσμια κρίση όμως θα πρέπει να ενισχύσουμε και την εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να υποστηρίξουμε τις προστάσεις του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία και το ελάχιστο κοινωνικό κατόφυλλο. Και μάλιστα τον Απρίλιο θα γίνει συνάντηση στην Ισπανία για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα, τα συναφή με τη στρατηγική του 2020. Και με τα συμπεράσματα αυτής της συνεδρίασης θα τροφοδοτηθεί η συζήτηση με νέα στοιχεία και θα δημιουργηθούν συνέργειε προκειμένου να εξέλθουμε από κοινού και συντονισμένα από την κρίση. Επίσης, ασχολούμαστε και με την ε, προετοιμασία της επόμενης ε, διάσκεψης κορυφής Υπουργών Απασχόλησης του G20 και εκεί θα υποβάλουμε προτάσεις για την επόμενη διάσκεψη κορυφής του G20 που θα γίνει στον Καναδά τον Ιούλιο. Η Ισπανική Προεδρία επιθυμεί στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα που κατά τη γνώμη μας είναι πρωταρχικά για την χάραξη της στρατηγικής του 2020. Χθε συναντήθηκα με τον ε, Επίτροπο και του έθεσα τους στόχους της Προεδρίας και πήρα από πρώτο χέρι κάποιες πληροφορίες για τις προτεραιότητες του υποψήφιου επιτρόπου. Η, η Ισπανική Προεδρία θα υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα ε, κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, η οδηγία για τη μητρότητα, για την τραυματισμό από αιχμηρά αντικείμενα, για την ε, ίση μεταχείριση των αυτόνομων αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων. Επίσης, ε, οι συμφωνίες σύνδεσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα της Προεδρίας και θα συνεργαστούμε για να προετοιμάσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε θέματα συντάξεων, νέων δυνατοτήτων για νέα θέσει απασχόλησης και άλλα θέματα κοινωνικο-εργασιακού ενδιαφέροντος. Όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στις διάφορες συνδιασκέψεις και οι μερίδες μελέτης που έχουν προβλεφθεί για το εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας και προσβλέπουμε και στη δική σας συμβολή και συνεργασία για τα θέματα αυτά. Εν κατακλείδη θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε τρεις τους ε, βασικούς στόχους της ε, Ισπανική Προεδρία σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων. Καταρχήν, συντονισμένη εργασία για την στρατηγική του 2020. Προώθηση από κοινού με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οδηγίε και νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Και τρίτον, πραγματοποίηση ενό χρονοδιαγράμματο ε, συνεδριάσεων που θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων για κέρια ζητήματα μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των κοινωνικών εταίρων. Θα ήθελα να σας αναγγείλω εν συντομία τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις που προβλέπονται. Στα πλαίσια της απασχόλησης, στη διάσκεψη για τις νέες ικανότητες, ε, δυνατότητες για το μέλλον της απασχόλησης, όπου θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί γνωστή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νέα προφίλ και τις νέες θέσεις απασχόλησης, θα γίνει στην Βαρκελόνη. Μία συνδιάσκεψη για τα κοινωνικο-εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων που θα γίνει στο Βιέδο. Τρει συνδιασκέψει ε, γύρω από τη δραστηριότητα των εργοδοτών και την αυτοαπασχόληση, αυτόνομη εργασία και κοινωνική οικονομία που θα γίνουν στη Σεβίλη, το Τολέδο και στην Πάλμα τη Μαγιόρκα. Και μία συνδιάσκεψη για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασία που θα γίνει στη Βαρκελόνη. Στα πλαίσια της κοινωνικής προστασίας θα διοργανωθεί μια συνδιάσκεψη για τις ελάχιστες συντάξεις και τη συμβολή του στην κοινωνική ένταξη. Αυτό θα γίνει στον Πούργος. Και σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση, μια υπουργική διάσκεψη ε, των Υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής και ε, Καραϊβική, στο Αλκαλά για την προώθηση τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Αυτέ ήταν συντομία οι προτεραιότητε τη Ισπανική Προεδρία σε θέματα απασχόληση και κοινωνική προστασία. Έχουμε ενώπιον μα μια πολύ σημαντική πρόκληση και αποστολή. Είμαστε υπέρ απρόσκοπτης ε, και διαφανούς συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και είμαι πρόθυμος και στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Έχω ήδη γεγραμμένους ε, ομιλητές που θέλουν να σας θέσουν ερωτήματα. Επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί προτίθεστε να συνεχίσετε το διάλογο και σας ευχαριστώ επίσης που εξ ονόματος της Επιτροπής μας ε, μας προσκαλέσατε στην διάσκεψη της Βαρκελόνης. Πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρης η παρουσίασή σας. Αλλά τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Τρινιδάδ Χιμένεθ, Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, για την πρώτη τοποθέτησή της. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Όπως και οι συνάδελφοί μου, ε, ο Υπουργό Απασχόληση και Υπουργό Ισότητα Ευκαιριών, χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα για τη σημερινή μου παρουσία στην Επιτροπή σα για να σα παρουσιάσω τι κατευθυντήριε γραμμέ και το πρόγραμμα τη Ισπανική Προεδρία σε θέματα κοινωνική πολιτική. Όπω ξέρετε, Ήδη αυτό το πρόγραμμα αποτελεί συμφωνία μεταξύ των τριών προεδριών, Ισπανικής, Βελγικής και Ουγγρικής, με βάση τις αρχές της υπευθυνότητας, της κοινή δράσης και της συνεργασίας. Θα ήθελα καταρχήν ε, να σας ε, πω μερικά λόγια για το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εκτιλήσεται η Ισπανική Προεδρία. Και από αυτό επηρεάστηκε και το πρόγραμμα εργασίας αυτή είναι η σοβαρότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική παγκόσμια κρίση που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο και ήταν πάρα πολύ σοβαρή και έδωσε έμφαση σε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Καταρχήν, η κρίση αυτή κατέδειξε την ε, ισχύ του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε ένα σύστημα οικουμενικής ευμάρειας με μια νομοθεσία που, θα, που είναι θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των πολιτών και με ένα σύστημα επαρκούς κοινωνικής προστασίας. Γύρω από αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετατράπηκε ε, το μοντέλο αυτό σε ένα σήμα κατά τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια πηγή έμπνευση και για πολλές άλλες χώρες λοιπόν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία σε όλες τις ε, στιγμές ε, της κρίσης και της οικονομικής δυσκολίας. Και αν μάθαμε κάτι από τις κρίσεις ε, του τελευταίου αιώνα είναι ότι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, η κοινωνική προστασία και η ενίσχυση των δικαιωμάτων είναι το μοντέλο που εξασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο την ευημερία. Είναι το μοναδικό μοντέλο που μπορεί να δημιουργήσει μια πιο δίκαιη κοινωνία και πιο ισότιμη κοινωνία. Η τελευταία κρίση λοιπόν έφερε στην επιφάνεια τον ευάλωτο χαρακτήρα πολλών στρωμάτων και ομάδων της κοινωνίας και κατέδειξε την ανάγκη, την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γι' αυτό και η στόχη αυτή... Ε, ε, ε, ήρθα στο προσκήνιο της, του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Προγράμματος. Μην ξεχνάτε, το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Αυτή η πραγματικότητα θα πρέπει να κατευθύνει όλες μας τις δράσεις, σε όλα τα επίπεδα, και στο εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας με πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να εξέλθουμε από την κρίση. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, η Ισπανική Προεδρία συμπίπτει με δύο ορόσημα, με δύο ιστορικές στιγμές που θα πρέπει να μετατρέψουμε σε ευκαιρίες. Καταρχήν, η Ισπανική Προεδρία συμπίπτει με τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, που διευρύνει τι εξουσίε τη Ένωση την, εμπλου, την εμπλουτίζει με νέα εργαλεία, νέους μηχανισμούς και ευκαιρίες, ενισχύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενισχύει τα θεσμικά όργανα, εκδημοκρατίζει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και δίνει περισσότερες ευκαιρίες δράσης, περισσότερους μηχανισμούς που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Επίσης, η Ισπανική Προεδρία συμπίπτει και με την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα και μετά το 2010. Θα πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια της οικονομίας της επόμενης δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ευρωβουλευτέ, χαράζουμε το μελλοντικό οικονομικό και πολιτικό κύκλο για την Ευρώπη μέχρι το 2020. Και στο πλαίσιο αυτό που σας παρουσίασα, η, η Ισπανική Προεδρία, ακούγοντας τις διάφορες χώρες και τους κοινωνικούς εταίρους, θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στα πλαίσια της μελλοντική μας στρατηγικής. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλουμε να αυξήσουμε την ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή μεταξύ των κοινοτικών χωρών, αλλά και μεταξύ των πολιτών μιας χώρας. Σε ό,τι αφορά τα θέματα κοινωνική προστασία, που είναι η δική μου αρμοδιότητα, η Ισπανική Προεδρία θα δώσει έμφαση στι ομάδε τη κοινωνία που είναι πλέον ευάλωτε. Για παράδειγμα, στους ε, ανθρώπους με αναπηρία, στους ηλικιωμένους και στις εθνικές μειονότητες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα στους τσιγκάνους, αθήγανους. Θα διοργανώσουμε λοιπόν ειδικέ υπουργικέ διασκέψει ε, με αντικείμενο την κατάσταση αυτών των ομάδων της κοινωνία. Θέλουμε αφενός να προωθήσουμε την ε, ένταξη αυτών που έχουν περισσότερε δυσκολίε πρόσβαση στην αγορά εργασία, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ε, μέρημνας ε, και σε θέματα υγείας για να καταργήσουμε τις ανισότητες. Επίσης, ε, θα δούμε τις σχέσεις μεταξύ των γενεών και το πρόβλημα της γύρασης του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεργαστούμε και με οργανώσεις αναπήρων για να χαράξουμε την στρατηγική μας για την επόμενη δεκαετία, γιατί τώρα θα χαράξουμε τους άξονες αυτής της στρατηγικής. Μας ενδιαφέρει η ευαισθησία, μας ενδιαφέρει όμως και η συμμετοχή, η προσωπική αυτονομία, η παιδεία και η απασχόληση. Θα προωθήσουμε τους κατάλληλους κοινωτικούς μηχανισμούς για να καταπολεμήσουμε τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Αθηγάνων που εξακολουθεί να ισχύει σε πολλές χώρες. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα θέλαμε να υποβάλουμε συμπεράσματα στο έπσκο του Ιουνίου για θέματα αναπηρίας, ε, γύρασης του πληθυσμού και διακριτικής μεταχείρισης βάρος των Αθηγάνων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανακήρυξη του 2010 ως του Ευρωπαϊκού Έτους ε, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και μάλιστα στις 21 έλαβε χώρα στη Μαδρίτη η εναρκτήρια σε διάσκεψη έγιναν τα εγγένεια αυτής της προσπάθειας με μια σημαντική ομιλία για το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης, μια ομιλία που έκανε ο Φελίπε Κονσάλες που είναι ο επικεφαλής ε, της ομάδας εργασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε και μια αξιολόγηση της, της στρατηγικής Λισαβόνας και τι έκανε αυτή για τη μείωση της φτώχειας στα διάφορα κράτη-μέλη. Έγινε επίσης μια ανάλυση των πιο σημαντικών εμπειριών, γιατί θέλουμε να μοιραστούμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Έγινε και μια στρογγυλή τράπεζα με μαρτυρίες ε, ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θέλουμε να ακούσουμε και τη δική τους φωνή για να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματά τους και σε αυτό το Ευρωπαϊκό έτος 2010 ε, κατά τις φτώχειες θα έχουμε την ένατη συνάντηση ε, ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας που θα γίνει τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας, εκπρόσωπος του οποίου βρέθηκε και στη Μαδρίτη. Η θεμελιώδη στόχη αυτού του Ευρωπαϊκού Έτου Καταπολέμηση Φτώχεια συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο με τι προτεραιότητε ε, του προγράμματο τη Ισπανική Προεδρία, αλλά και με τι ε, αρχέ τη Ευρωπαϊκή Προεδρία. Καταρχήν, η καινοτομία είναι σημαντική προτεραιότητα. Και όταν λέω καινοτομία, δεν εννοώ μόνο την τεχνολογική, αλλά και την οικονομική και τη θεσμική και την πολιτική. Όλε αυτέ οι καινοτομίε θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και να εμβαθύνουμε στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την ισότητα ανδρών και γυναικών, την αλληλεγγύη και την αναπτυξιακή βοήθεια. Η Ευρώπη που έχουμε κατά νου είναι μια καινοτόμα πρωτοπόρα φιλόδοξη Ευρώπη, προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις με θεμελιώδη αξία την ισότητα, την ευημερία και την ισότητα ευκαιριών. Το 2010 λοιπόν κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτέ θα είναι ένα καλό έτος για να διατρανώσουμε τις αρχές και τους στόχους μας και να προβλέψουμε τα απαραίτητα μέσα για να τους υλοποιήσουμε. Θα είναι καλό έτος γιατί θα γίνει μια αναθεώρηση της στρατηγικής Λισαβόνας και θα περάσουμε σε ένα νέο κύκλο κοινωνικού προγράμματος και Προσβλέπουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη στρατηγική του 2020, αλλά και για τη διαμόρφωση ενός ε, νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προγράμματος, αν το αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προτείνει στο επόμενο εξάμεινο. Φυσικά προσβλέπουμε και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα έχει νέο, ανανεωμένο και ενισχυμένο ρόλο χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να έχει κέρια θέση στη συζήτηση. Η Ισπανική Προεδρία ε, έχει επίγνωση των χαλεπών καιρών και των προκλήσεων και γι' αυτό έχει ε, αναγάγει την εμβάθυνση στην κοινωνική Ευρώπη σε ύψιστη προτεραιότητα μαζί με την προώθηση του νέου οικονομικού μοντέλου που θα μας επιτρέψει να εξέλθουμε από την κρίση ανακτώντας όμως τις θέσεις απασχόλησης που χάσαμε. Και φυσικά περιμένουμε τη συμβολή σα και τη συνεργασία σα για να διεκπαιρεώσουμε το φιλόδοξό μα πρόγραμμα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ε, το θεσμικό όργανο με τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία, που βρίσκεται πιο κοντά στου πολίτε και σε αυτέ τι κοινωνικέ ομάδε τι πιο ευάλωτε. Και η Ισπανική Προεδρία είναι απόλυτα ανοιχτή και πρόθυμη για το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με προσήλωση θεσμική και αφοσίωση στη συνεργασία. Και όπω είπε και ο συνάδελφο Υπουργό Απασχόληση. Είμαι και εγώ στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε για την διαθεσιμότητα που δείχνετε και βεβαίως σας ευχαριστούμε ε, που θα ξεκινήσει μια συζήτηση βάσει των λεγόμενων σας. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βιβιάννα Αίδο, Υπουργό Ισότητας των Φίλων, για να παρουσιάσει και εκείνη τις ιδέες της. Και παρεμπιπτόντως να πω ότι κλείνει ο κατάλογος των αγορητών. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι και εγώ ιδιαίτερη τιμή για την παρουσία μου στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων μαζί με τους ε, συναδέλφους, τον Υπουργό Απασχόλησης και την ε, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Ε, οι τρεις μας θα προεδρεύσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ αυτό το εξάμεινο. Ήδη έκανα την ομιλία μου στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναίκας και ισότητα των Φύλων και μίλησα για την ανάγκη προώθηση ε, της πολιτικής ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό θα είναι ο μύτος της Αριάδνης του προγράμματος της Προεδρία Προεδρίας που θα ασκήσει την Προεδρία αυτή στο πρώτο εξάμεινο του 2010. Θέλουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και έναν προγραμματισμό για την επόμενη δεκαετία. Η ισότητα είναι αναφυσβήτητα ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι θεμελιώδης δικαίωμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Η ισότητα όμως είναι θέμα και αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας. Δύο παράγοντες διαμορφώνουν την πρόκληση Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό και τη χάραξη κοινών πολιτικών. Ο ένας παράγον είναι η βαθύτατη οικονομική κρίση η ε, πιο σοβαρή των τελευταίων δεκαετιών, από την οποία αρχίζουμε και ξεφεύγουμε. Και το ο δεύτερος παράγοντας είναι η χάραξη μιας νέας οικονομικής στρατηγικής ανάκαμψης με χρονικό ορίζοντα το 2020. Και τα δύο αυτά θέματα θα αποκτήσουν κέρια σημασία στο Ισπανικό εξάμεινο. Ξεκινούμε από τη βάση της στρατηγικής της Λισαβόνας και από τους προσανατολισμούς αυτούς, γιατί δεν έχουμε υλοποιήσει πλήρως τους στόχους της Λισαβόνας. Αλλά δεν είναι λογικό να απομακρυνθούμε από το μονοπάτι αυτό, μια και βασική στόχη ήταν η ισότητα ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Και για να υλοποιήσουμε ένα μοντέλο κοινωνική αηφορία και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το ταλέντο και το δυναμικό που έχουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν το 59% των ανθρώπων που είχαν πτυχίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2006. Είναι οι περισσότερες ε, απόφυτοι, ανώτατο σχολό και παρόλα αυτά έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και η στρατηγή του 2020 θα πρέπει να διευρύνει τους στόχους υπέρβασης των κοινωνικών προσκομμάτων ε, και αυτής της αδικίας που οδηγεί και σε μια οικονομική δισκαμψία. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα της Σουηδική Προεδρία στο τελευταίο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του 2009. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Θα πρέπει να διευκολύνουμε αυτή την αλλαγή προκειμένου να γίνει ένας πιο ισότιμος καταμερισμός των καθηκόντων στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο. Γιατί η ανατροφή των παιδιών και ο οικογενειακό βίος δεν είναι ίδιο και προνόμιο το γυναικό. Θα πρέπει να γίνει καλύτερος καταμερισμός των ε, οικογενειακών βαρών και επίσης ε, να προωθήσουμε την καλύτερη φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων στην οικογένεια, κυρίως αυτών που είναι από 0 έως 3 ετών. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα και να υλοποιήσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Βαρκελόνης του 2002. Έχουμε φυσικά και την πρόταση οδηγία για την μητρότητα για την οποία θα κληθείτε να καταρτήσετε και γνωμοδότηση. Είμαστε υπέρ μιας πρότασης που θα προστατεύσει την υγεία και τα δικαιώματα της εργαζόμενης γυναίκας, ε, που είτε είναι έγκυος, είτε λεχόνα, είτε γαλουχούσα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν θετικά στην υγεία της μητέρας, θα πρέπει να βοηθήσουν την σωματική της ανάνυψη και ταυτόχρονα να αυξήσουν την ε, ασφάλεια δικαίου και τα εχέγγυα πρόσβαση στην αγορά εργασία και να διευκολύνουν και τη συμφιλίωση της επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Και όλα αυτά δίνοντα έμφαση στη συνυπευθυνότητα. Δυστυχώ υπάρχουν τεράστιε μισθολογικέ διαφορέ, ένα πραγματικό μισθολογικό χάσμα που αποτελεί μια αφόρητη διάκριση ει βάρο των γυναικών που παρεμποδίζει την επαγγελματική του ολοκλήρωση. Γι' αυτό και χρειάζονται κάποιοι κρατικοί μηχανισμοί, αλλά και κάποια διαπαιδαγώγηση και να πεταχθούν αυτές οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα των δύο φύλων που κρατάει κλειστού ορισμένου κλάδους στις γυναίκες. Θα πρέπει να διαταράξουμε αυτή την αδράνεια και αυτή τη διακριτική μεταχείριση που αποβαίνει βάρο τη κοινωνία. Επίση, θα πρέπει να προωθήσουμε την συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικέ θέσει σε ηθήνουσες θέσεις και σε λήψη αποφάσεων για να συμμετέχουν καλύτερα οι γυναίκες σε αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Με παρόμοια επίπεδα κατάρτισης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Αυτό θα πρέπει να το αντιστρέψουμε και στην άτυπη διάσκεψη κορυφή Υπουργών Απασχο... Ε, Ισότητας που θα γίνει στη Βαλένση 25 και 26 Μαρτίου θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε το ρόλο των πολιτικών ισότητες στο ισχύον οικονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι σημαντική προτεραιότητα της ε, Ισπανικής Προεδρίας, όπως και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μάλιστα, επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο συμπερασμάτων που ευελπιστούμε ότι θα εγκριθούν στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, που θα γίνει 8 και 9 Μαρτίου. Εκεί αναφέρον, αναφέρεται η πρόταση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών, την θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, για τα θύματα τέτοιας βίας και την ε, θέσπιση μιας ενιαίας ε, πράσινης γραμμής για τα θύματα της βίας των φύλων. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση άσχετα από το που οφείλεται και αναφέρομαι στην οδηγία για την ίση μεταχείριση. Θα ήθελα ολοκληρώνοντα, κυρίε και κύριοι, να σα υπενθυμίσω ότι η ισότητα ποτέ δεν ήταν πρόβλημα τη Ευρώπη. Το αντίθετο. Η ισότητα ήταν ανέκαθεν παράγων κοινωνικής πρόοδου και οικονομικής ανάπτυξης. Σήμερα όμως, περισσότερο από ποτέ, η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί τμήμα της λύσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί πλήρω στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την υλοποίηση ισότιμου και ανταγωνιστικού κοινωνικού μοντέλου, στο οποίο προσβλέπουμε όλοι. Σα ευχαριστώ θερμά και όπω και οι συνάδελφοι, είμαι στη διάθεσή σα για τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Nous allons... Euh, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ε, ερωτήσεις και για να μην ξεφύγουν οι υπουργοί ε, θα ε, παίρνουμε τις ερωτήσεις 4-4. Ο κύριος Αλεσάνδρος Θέρκας και μετά η κυρία Σρέτερ. Κύριε Θέρκας παρακαλώ. Και ε, βεβαίω ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά πράγματα να πείτε, αλλά θα ήθελα να μην μακρηγορήσετε παρακαλώ πολύ. Así Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και τις δύο γυναίκες υπουργού. Έχουμε υψηλές προσδοκίες από την Ισπανική Προεδρία. Χαιρετίζουμε τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση και την προσήλωση που δείξετε στα εργατικά δικαιώματα, στην κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις πολιτικές ισότητες. Και έχω μία ερώτηση για τον καθένα από εσά. Κύριε Υπουργέ Κορμπάτσο, τη στιγμή που υπάρχει ένας προφανής πειρασμός σε αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση να συρρυκνωθεί η κοινωνική προστασία των εργαζομένων για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Μας ανησυχεί αυτή η τάση του Συμβουλίου που φάνηκε και στη συζήτηση για την οδηγία της απόσπασης των εργαζομένων. Γιατί εκεί ε, θέλουν από την Κερκόπορτα να επαναφέρουν την οδηγία Μπόλκεστάν και να ισχύσουν οι λιγότερο ευμενείς κανόνες της ε, χώρας ή έχουμε και την οδηγία για το ωράριο εργασία που θέλουν να μα επαναφέρουν στο 19ο αιώνα και στι βιομηχανικέ σχέσει που επικρατούσαν τότε με τεράστια κοινωνική ανασφάλεια. τι θέση έχουν ε, τα εργατικά δικαιώματα σε μια περίοδο κρίση, κύριε Υπουργέ. Κύριε Χιμένε, ξέρω πόσο προσιλωμένη στο θέμα της δημόσιας υγείας και πόσο προωθήσατε την οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Το θέμα είναι όμως ότι τα υγειονομικά συστήματα σχετίζονται και με τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί τον τελευταίο αιώνα. Πώς ε, ε θα προσπαθήσετε να άρετε τη σύγκρουση μεταξύ του κανονισμού 1408 και της νέας οδηγίας. Γιατί δυστυχώς ε, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ε, έρχονται αντιμέτωπα με μια πολύ γενναιόδορη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μάλλον όμως θα είναι ανέφικτη. Κυρία Ίντο, ξέρουμε το τεράστιο έργο σας για θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών και παρόλο που αρχίζουμε και γερνάμε, ε, μην μας ξεχνάτε στα θέματα της ισότητας ή τους πιο ηλικιωμένου ή όσους έχουν κάποια αναπηρία, γιατί και αυτοί καλύπτονται μερικές φορές από ή υφίστανται την διακριτική μεταχείριση. Μιλήσατε για το μισθολογικό χάσμα και για τη μητρότητα. Πώς θα φροντίσετε όμως στο Συμβούλιο να περάσει αυτή η θεσπέσια μουσική υπέρ της μητρότητας σε πιο απτά αποτελέσματα και δράσεις. Ευχαριστώ κυρία Σρέντερ και μετά κύριο Σκομφεράτη. Ευχαριστώ. Δύο ζητήματα με ενδιαφέρον. Καταρχάς μιλήσατε για τις προτεραιότητες σας το πρώτο αυτό εξάμεινο. Εμένα με, ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει εάν θα πιέσετε την Κομισιόν να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ή θα κινηθείτε μέσα στον κοινωνικό διάλογο. Ε, μου είπατε ότι θα οργανώσετε και ένα συνέδριο με θέμα την ε, ένα συνέδριο εργασίας δηλαδή για να συζητήσετε το θέμα αυτό και είπατε ότι στη Βαρκελόνη θα οργανώσετε ένα συνέδριο για νέους τομείς εργασίας. Με ενδιαφέρει ποιος είναι ο στόχος αυτού του συνεδρίου και τι σκοπεύετε να κάνετε στο θέμα των νέων τρόπων, νέων εργασιών. Ευχαριστώ πολύ. Σάρζο Κονφεράτη και μετά ο κύριο Τσεμπάουε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον το πλαίσιο ε, το οποίο μας παρουσίασαν οι φιλοξενούμενοι μας και πιστεύω ότι η κοινή εργασία τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ότι ε, έχουμε εδώ εκπροσώπους τριών διαφορετικών Υπουργείων που όμως καθημερινά συνεργάζονται. Ε, είναι πραγματικά, είναι λέγω, μια πολύ θετική ε, προσέγγιση την οποία συμμεριζόμαστε απόλυτα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους φιλοξενούμενους μας να μας δώσουν, αν είναι σε θέση, κάποια λεπτομεριακά στοιχεία όσον αφορά τα τρία θέματα τα οποία μας απασχολούν. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε για ανεργία ε, και γιατί η ανάκαμψη από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι τέτοια που να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Επομένως, ε, ακόμα υπολείπεται χρονικό διάστημα στο οποίο θα αυξάνεται η ανεργία. Ανεργία η οποία πλήγει, πλήττει περισσότερο τους νέους, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά οι οποίοι θα μείνουν ακόμα έξω από την αγορά εργασίας. Ε, ερωτώ λοιπόν, στις προθέσεις σας περιλαμβάνονται ε, πρωτοβουλίες ε, οι οποίες θα αφορούν την ανεργία των νέων. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τη γύρανση. Βεβαίως υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, ενώ από την άλλη πλευρά το προσδόκιμο ζωής μεγαλώνει. Ε, ευτυχώς ζούμε περισσότερο, δυστυχώς γεννιούνται λιγότερα παιδιά, επομένως το κοινωνικό βάρος το οποίο προκύπτει είναι σημαντικό. Άρα θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν σχετικά και με την προστασία των ηλικιωμένων ε, προβλέπεται κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Τρίτον, για να διατηρηθεί η αγορά εργασίας και επομένως και η, παραγωγικότητα της Ευρώπης. Θα πρέπει να βασιστούμε και σε ξένους, σε ανθρώπους εργαζόμενους που έρχονται από άλλες χώρες. Αυτό όμως προϋποθέτει η ικανοποιητική, συγγνώμη, ικανοποιητικό έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να ζήσουν καλά μαζί μας έτσι ώστε να οικοδομήσουμε το μέλλον. Όμως θα πρέπει να θίξουμε το θέμα της ένταξης, της ενσωμάτωσης των ανθρώπων αυτών. Μπορείτε να μας πείτε κάτι και προχωρώντας παραπέρα ακόμα και για το ζήτημα της ηθαγένειας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής αυτής της πρώτης ομάδας, ο κύριος Σαμπάουι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα η στρατηγική του 2020. Σε αυτήν την στρατηγική δεν έχουμε ακόμα πολλά απτά συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε κάποιες σφαιρικές ε, και μάλλον ασαφείς ιδέες. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την στρατηγική 2020. Πολύ θα με ενδιέφερε να ακούσω εάν προτίθεστε να δημιουργήσετε ε, εγγυήσει, ε, να δώσετε κάποια εχέγγυα. Γιατί έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την εγγύηση υλοποίησης, γιατί και στη Λισαβόνα λέγαμε πολλά ωραία, αλλά δεν καταφέραμε ε, να τα υλοποιήσουμε και μάλιστα δεν ξέρουμε μέχρι ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Επίσης, υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στη στρατηγική 2020 και τις πολιτικές συνοχής, γιατί δεν έχει γίνει αναφορά σε αυτή την διασύνδεση ανάμεσα στις δύο τόσο σημαντικές πολιτικές. Ε, επίσης έγινε λόγος για ένα τρίο προεδρίας, πράγμα που σημαίνει ότι η Ισπανική Προεδρία θα συνεργαστεί με την Βελγική και την Ουγγρική Προεδρία. Ε, νομίζετε ότι αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε ότι θα, θα μπορέσετε να λύσετε κάποια ε, προβλήματα, κάποια τα οποία θα αφήσετε ενδεχομένως... Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω επιγραμματικά. Για το θέμα της οδηγίας για το ωράριο εργασίας. Γνωρίζουμε όλη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωρίζουμε τη θέση του Συμβουλίου και περιμένουμε τις εξελίξεις. Η Ισπανική Προεδρία πάντως θα υποστηρίξει την προηγούμενη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Η Ισπανική Προεδρία θα προσπαθήσει να προωθήσει μια έξοδο από την αποτελμάτωση, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πρώτα απ' όλα την αρχή ίση αμοιβή για ίση εργασία. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι ε, η βασική αρχή που θα, μα, θα μας εμπνέει και στο μέλλον. Αναφέρθηκε και το θέμα της συνδιάσκεψης που θα γίνει στο, στο Οβιέδο για την οδηγία, για την απόσπαση εργαζομένων. Στις σημερινές μελέτες που θα γίνουν στο, στο Οβιέδο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου, των κρατών μελών, ελπίζω να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμπειρογνώμονε και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Στόχο τη διάσκεψη αυτή είναι να γίνει μια διεξοδική ανάλυση και να αντληθούν κάποια συμπεράσματα για να δοθεί μια όθηση στην ε, περαιτέρω συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τη συνδιάσκεψη για τι νέε θέσει απασχόληση, η συνδιάσκεψη αυτή προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενδιαφέρεται για τη συζήτηση αυτή για τις νέες μορφές εργασίας, για τα νέα προφίλ, τα νέα χαρακτηριστικά και εκεί φυσικά θα συμμετέχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Ισπανική Προεδρία και ε, θα εμπλουτιστεί η συζήτηση. Μια άλλη ερώτηση που τέθηκε ήταν ε, πολύ ουσιαστική και έθεσε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Η Ευρώπη χάραξε μια στρατηγική για το 2010 που δυστυχώς δεν κατάφερε να υλοποιήσει εξαιτία της οικονομικής κρίσης. Τώρα καλείται να χαράξει μια νέα στρατηγική μέχρι το 2020 και κατά τη γνώμη μου θα ήταν λάθος να αγνοήσουμε την πραγματικότητα και να ξεχάσουμε την παρούσα συγκυρία ή το μακροπρόθεσμο. Χρειαζόμαστε μία διπλή προσέγγιση. Μία προσέγγιση ως προς τη συγκυρία που θα λαμβάνει υπόψη τη συγκυρία και θα δίνει μια απάντηση στους νέους και στην απασχόληση, αλλά χρειαζόμαστε και μια μεγαλύτερη διορατικότητα και ένα πιο μακρόπνο και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Σίγουρα η γύραση του πληθυσμού έχει και κοινωνικές επιπτώσεις. Βέβαια, στις δικές μου αρμοδιότητες σχετίζεται περισσότερο με το θέμα των συντάξεων. Και η Ισπανική Προεδρία θα διοργανώσει διάσκεψη για την κινητικότητα, τις συντάξεις ε, με προοπτική το 2030-2040. Γιατί τότε το παθητικό δυναμικό θα έχει διπλασιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να επινοήσουμε νέα μέτρα για να διασφαλίσουμε το κράτος πρόνοιας και ευημερίας. Το θέμα της μετανάστευσης. έχει σταματήσει προ το παρόν η οικονομική μετανάστευση, αλλά όταν ξεφύγουμε από την κρίση θα χρειαστούμε περισσότερου οικονομικού μετανάστε. Επίση, έχουμε μια πρόταση οδηγία για την ενιαία άδεια που εναρμονίζει τι συνθήκε για όσου έρχονται νόμιμα για να εργαστούν στην Ευρώπη. Αυτή την οδηγία θα επεξεργαστούμε ε, και βρίσκεται σε φάση πρώτη ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της στρατηγικής για το 2020. Βρισκόμαστε σε φάση προβληματισμού και ανάλυσης αυτής της στρατηγικής. Η Ισπανική Προεδρία θα προλειάνει το έδαφος ώστε στο Ερεινό Συμβούλιο να αποκρισταλωθεί κάποια θέση για τη στρατηγική του 2020 που είναι στόχος, αναγκαιότητα και θα χρειαστούν οι ανακοινώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλουμε όμω η στρατηγική του 2020 να είναι διαφορετική από τη στρατηγική τη Λισαβόνα, θα πρέπει η στρατηγική του 2020 να μην περιορίζεται μόνο σε φιλοσοφικές διακήρυξεις αξιών, αλλά και σε αυτά προγράμματα αξιολόγησης, συντονισμού και διακυβέρνησης. Αλλιώς θα διατρέξουμε τον κίνδυνο να γίνει γνωστή η στρατηγική του 2020 στους συμμέτερους, στα θεσμικά όργανα, στους εμπειρογνώμονες, αλλά να βρει παγερά αδιάφορους τους πολίτες και να μην τους ξυπνήσει κανένα ενδιαφέρον θα πρέπει οι πολιτικοί να μην μένουν μακριά από το πολίτη και να μην χρησιμοποιούν μια τεχνοκρατική ξύλινη διατύπωση που δεν θα αγγίζει τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα πρέπει να βρεθούμε κοντά του και να τον αγγίξουμε τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποια από τις δύο κυρίες Υπουργούς να απαντήσει. Παρακαλώ ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση για τα δικαιώματα υγείας, τα υγειονομικά δικαιώματα και την κινητικότητα των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα και στην τελευταία υπουργική διάσκεψη, παρόλο που καταλήξαμε σε συμφωνία για το περιεχόμενο της οδηγίας, η Ισπανική Προεδρία ήταν έτοιμη να αναστήσει ευρύτερη συνένεση ως προς πιο φιλόδοξους στόχους για να υλοποιήσουμε τα δικαιώματα των ασθενών και την εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών ώστε να υπάρχει καταρχήν ένας ιατρικός λόγος για την κινητικότητα, να επιβεβαιώνεται Επίσης θα πρέπει τα κέντρα περίθαλψης να εντάσσονται σε ένα δημόσιο κρατικό σύστημα ή και αν, είναι, αν ανήκουν στον ιδιωτικό κλάδο να υπάρχει κάποιος συντονισμό. Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη κυρίες και κύριοι είναι ότι ίσως υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις και άρα να μην υπάρχει ασφάλεια δικαίου γιατί οι κανονισμοί ασχολούνται με το θέμα της κινητικότητας αλλά επεξεργαζόμαστε μια οδηγία που πολλές φορές έρχεται σε αντίφαση με τους κανονισμούς. Με τον κανονισμό μάλλον. Ο κανονισμός 883 του 2004 που θα τεθεί σε ισχύ μόνο φέτος το 2010 μετά την έγκριση και των ε, ε εκτελεστικών κανονισμών 987 και 988 του 2009 ε, ανταποκρίνεται και στην ομολογία του ΔΕΚ. Για παράδειγμα, δίνει μια απάντηση στις, στις λίστες αναμονής. Στο άρθρο 20 του 883 δίνει δικαίωμα περίθαλψης όταν ε, βρίσκεται σε μια εκτενή λίστα αναμονή στο κράτο προέλευση να μπορεί να τύχει περίθαλψη αλλού. Επίση, μιλάει για τι προσωρινέ παραμονέ σε άλλε χώρε. Γίνεται επιστοποίηση δικαίου μέσω της, ε, του Ευρωπαϊκού Βιβλιαρίου Υγείας. Το άρθρο 19 του κανονισμού 883 δίνει απάντηση σε θέματα παραμονής ε, σε άλλο κράτος ε, που δεν είναι το αρμόδιο και επίσης δίνει απάντηση στις προγραμματισμένες θεραπείες που προϋποθέτουν άδεια, προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης, ε, μιλάει για κάποια διασυνοριακά ζητήματα. Ο κανονισμός 1408 δεν περιλάμβανε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να προτείνουμε οδηγία. Ο κανονισμός 883 στα άρθρα 17 και 18 προβλέπει ότι αν τεθούν σε ισχύ οι εφαρμοστικοί κανονισμοί, η περίθαλψη των ασθενών που βρίσκονται σε παραμεθόρειες περιοχές να καλύπτεται από τον κανονισμό. Πάντως ε, συνεργαζόμαστε και με την, Ισπανία, και με την Πορτογαλία και με τη Γαλλία και έχουμε διάφορες συμφωνίες. Η προσπάθειά μας πάντως θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση ευρωπαϊκής λύσης προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα πακέτο υγειονομικής περίθαλψης και παροχής που θα είναι κοινό σε όλες τις χώρες και που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών και θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μας. Θέλουμε μια φιλόδοξη λύση που θα είναι συμβατή με τους κανονισμούς και που θα δίνει πραγματική λύση στα προβλήματα των ασθενών που έχουν επισημάνει και η νομολογία του ΔΕΚ αλλά και οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό θα είναι το επικοδομητικό πνεύμα που θέλει να υιοθετήσει η Ισπανική Προεδρία για το θέμα αυτό και λυπούμε που μακρηγόρησα κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ εν συντομία να απαντήσω σε δύο ερωτήσει. Κύριε Σέρκας, θέλουμε πρώτα απ' όλα να πείσουμε, όχι να κατανικήσουμε. Και για να πείσουμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της λογικής. Είναι αδύνατο να, να αγνοούμε τις γυναίκες. Είναι κρίμα να μην αξιοποιούμε το τεράστιο δυναμικό τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα τους. Είναι πραγματικά μια σπατάλη αυτό και δεν έχουμε την πολυτέλεια μιας τέτοια σπατάλης. Οι γυναίκες είναι πάνω από το μισό του πληθυσμού και έχουν τεράστιες ικανότητε. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ισότητα όχι για θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για την πιο αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων πόρων. Και αν θέλουμε να υπάρξει συνένεση ότι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο θα στηρίζεται στην αηφορία, αηφορία δεν νοείται μόνο υπό το πρίσμα το περιβαλλοντικό ή το οικονομικό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την κοινωνική βιωσιμότητα και την κοινωνική αηφορία που έχει ως άξονα δράσης τον άνθρωπο. Θα είναι ανθρωποκεντρικό αυτό το μοντέλο, όχι όπως ε, το ολέθριο μοντέλο που μας οδήγησε στην καταστροφή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και θα πρέπει να υπολογίζουμε σε όλους τους πολίτες και στις γυναίκες. Και η στρατηγική του 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διάσταση της ισότητας των φύλων και τη, της του μισθολογικού χάσματο τη αύξησης τη απασχόλησης των γυναικών θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη συνυπευθυνότητα και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο χώρο, στον καλύτερο καταμερισμό των οικογενειακών βαρών, στην ε, ε, συμμετοχή, καλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία μεταξύ τη της των 53 και 60 ετών, γιατί εκεί το ποσοστό απασχόληση είναι μόνο 39%. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, προσπελάσιμες υπηρεσίες φροντίδας και να προωθήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών σε ηθήνουσες και ηγετικές θέσεις. Αυτή είναι η στόχη της Ισπανικής Προεδρίας και ελπίζω να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτά. Σε ό,τι αφορά τη μία της οδηγίας για την ίση μεταχείριση, όντως θέλουμε να γίνει μια εναρμόνιση του επίπεδου προστασίας ε, έναντι οποιασδήποτε μορφής διακριτικής μεταχείρισης για αναπηρία, ε, γενετήσιο προσανατολισμό, ηλικία, θρησκεία, κτλ. Ήδη είχαμε μια οδηγία για την ισότητα της μεταχείρισης πέραν του εργασιακού χώρου και προτείναμε οδηγία για καταπολέμηση της διάκρισης για λόγους ε, φύλου ή άλλων αιτίων. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, ε, να προλιάνουμε το έδαφος και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για συνένεση Υπάρχουν επιφυλάξει από ορισμένα κράτη-μέλη. Πάντω ήταν απογοητευτικό να μην καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατοχυρώσει μια ελάχιστη μορφή προστασία εναντί οποιασδήποτε μορφή διακριτική μεταχείριση. Άλλωστε κάτι τέτοιο προβλέπεται και στην ίδια τη συνθήκη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσει ο δεύτερο γύρος των ε, αγορητών. Ε, θα ζητήσω από του ομιλητέ να απευθύνουν συγκεκριμένη ερώτηση σε συγκεκριμένο ε, υπουργό και όχι 15 ερωτήσει. Ε, μία ερώτηση ο καθένας. Κυρία Λίν πρώτα. Uh, έχω δύο ερωτήσεις. Όσον αφορά το χρόνο, την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, χαίρομαι ιδιαίτερα που στην Επιτροπή μας θα προχωρήσουμε το θέμα της ε, συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για το... possibility of... Αλλά τώρα όσον αφορά ε, το διαχωρισμό από τον τομέα της υγείας, ήθελα να ρωτήσω την Ισπανική Προεδρία πιστεύετε ότι θα επιτύχετε μια συμφωνία για την οδηγία του χρόνου εργασίας, ότι θα το καταφέρετε αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση αποφορά την αποφυγή και πρόληψη των διακρίσεων στις, προς τις δύο κυρίες υπουργού. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρετε την οδηγία κατά των διακρίσεων και την ε, βούλησή σας να την προωθήσετε. Ε, μπορείτε να μας ενημερώσετε αν έχετε ξεκινήσει προκαταρτικές συζητήσεις, πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στις διαβουλεύσεις και αν πιστεύετε ότι η εξάμεινη ε, Προεδρία ε, αρκεί για να ολοκληρώσετε το φάκελο αυτό. Η τρίτη ερώτηση αφορά την κονιακή βία. Όταν το παρατηρητήριο ιδρύθηκε, ή θα θα ιδρυθεί, θα εξετάσει την κονιακή βία εναντίον ανδρών όπως και, κατα... και εναντίον γυναικών. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου και οι άνδρες υπήρξαν θύματα οικογενειακής βίας και δεν θα ήθελα να εστιάσουμε το θέμα αυτό μόνο στις γυναίκες. Ε, αυτό θα με δυσαρεστούσε ιδιαίτερα. Ε, πολλές φορές υπάρχουν ε, πραγματικά ε, τρομερά, τρομερή βία κατά των ανδρών, η οποία δεν αναφέρεται. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις υπουργούς για την παρουσίασή τους ε, του προγράμματος της Ισπανικής Προεδρίας. Είναι πολύ σημαντικά όλα τα θέματα αυτά για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εύχομαι μια καρποφόρο θητεία. Ε, καταρχάς προς τον Υπουργό κύριο Καρμπάτσιο. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Διότι εάν δεν ληφθούν ε, μέτρα, ειδικά μέτρα για τους νέους, η Ευρώπη θα χάσει το τρένο, όπως λέμε. Ε, τι μέτρα λοιπόν έχουν υπόψη τους να λάβουν για να διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των νέων ανθρώπων και δι' των νέων που εισέρχονται ή επισημούν να εισέλθουν στην αγορά εργασία πρώτη φορά. Εν συνεχεία προς την κυρία Υπουργό Χιμένες. Υπάρχουν 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σήμερα περίπου που ζουν κάτω από το επίπεδο της στόχιας και αγωνίζονται με, υπό τις παρούσες συνθήκες της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Τι μέτρα λοιπόν θα λάβετε για να παγιώσετε ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορέσει ε, να είναι αποδέκτης των βασικών κοινωνικών επιδομάτων. Τι μέτρα θα λάβετε για να μπορέσετε να ανυψώσετε, να αναβαθμίσετε το κοινωνικό τους επίπεδο στην Ευρώπη και προς την Υπουργό κυρία Ιντό. Ε, έχουμε τώρα την στρατηγική του 2020 και ένας από τους στόχους είναι η καταπολέμηση των εκκρίσεων κατά των γενικών και δι κατά των εγγύων γαλουχουσών και λεχόνων γυναικών ε, στο χώρο εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι μέτρα θα λάβετε όσον αφορά την εργασιακή ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ποια μακροχρόνια μέτρα θα λάβετε λοιπόν για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση της ανισότητας και των διακρίσεων μεταξύ των φίλων. Ο κύριος ε, Καζα... Ε, Κοζά, πρώτος ομιλητής. Ε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που διαπιστώνω ότι η, χρήση, η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ξαναμπαίνει στις προτεραιότητες ε, και εδώ βλέπουμε ε, ότι ο αριθμός ε, είναι πολύ σημαντικός. Το τρίο της Προεδρίας έχει δεχτεί ότι υπάρχουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία οι οποίοι θέλουν να απασχοληθούν. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς θα διασφαλίσετε την αύξηση του ποσοστού απασχολησιμότητας των αναπήρων, των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, έχετε πρωτοβουλίες, προβλέπετε πρωτοβουλίες ε, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για περισσότερες θέσεις εργασίας δεν ξέρω ποιος από τους τρεις υπουργούς ε, θα απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ε, επίσης, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προετοιμασία της οδηγίας για την άρση των, της διακριτικής μεταχείρισης. Γνωρίζομαι ότι η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά την άρση τέτοιων εμποδίων ε, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση ε, σχετικά ε, με την προσβασιμότητα προς ε, όλες ε, τις ε, υπηρεσίες και όλες τις πρωτοβουλίες και εγώ θα ήθελα να ζητήσω το χρονικό περιθώριο για την άρση όλων των εμποδίων να είναι τα 10 χρόνια και όχι τα 20. Άτομα με αναπηρία, αθήγανοι, μειονοτικές ομάδες, τι θα κάνετε συγκεκριμένα έτσι ώστε να λύσετε τα προβλήματα πρόσβαση στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία ε, Υπουργέ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις αποφεύγοντας την επανάληψη. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική 2020, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ε, και ανησυχίες για την ανεργία των νέων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασε το 21% αυτή η ανεργία των νέων. Ε, Υπουργός Χιμένες μίλησε για κάποια απτά μέτρα για τις εθνικές μειονότητες. Οι νέοι, οι μετανάστες, οι από εθνικές μειονότητες ε, μαστίζονται από πολύ υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους υπόλοιπους νέους στην Ευρώπη. Θα λάβετε σε αυτό το εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας ε, κάποια μέτρα θα προτείνετε κάποια μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση των νέων που είτε είναι μετανάστες είτε προέρχονται από εθνικές μειονότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, la primera... Ευχαριστώ. Τέθηκαν ερωτήσεις ε, για την οδηγία του ωραρίου εργασίας. Με ρωτήσατε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, πώς θα επιδιωχθούν συμφωνίες και αν θα μπορούσε να, αποκλειστεί, να διαχωριστεί ένας ε, συγκεκριμένος κλάδος όπως της υγείας. Η Ισπανική Προεδρία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την ε, σύναψη συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κοινωνικών Εταίρων. Ελπίζουμε, χάρη στο διάλογο, να καταλήξουμε σε συνένεση και σε μια οδηγία που θα τύχει της υποστήριξης όλων των θεσμικών οργάνων. Πάντως, το θέμα της πιθανότητας υλοποίησης στην οδηγία ενός συγκεκριμένου θέματος, του αποκλεισμού του κλάδου υγείας, για παράδειγμα, όπως προτάθηκε. Αν προτεραιότητα, προτεραιότητά μα έχουμε το γενικό και μόνο σε περίπτωση απο, αποτυχίας στα γενικά θα ασχοληθούμε με πιο ειδικά ζητήματα, με ειδικού κλάδους. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανεργίας των νέων, το θέμα είναι επίγον να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Γιατί το πρόβλημα αυτό είναι εγκάρσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών, αλλά το πρόβλημα είναι κοινό. Και στην πρώτη γραμμή του πυρός βρίσκονται οι νέοι, είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία. Ω προ τη διάγνωση συμφωνούμε. Αν όμω δεν λάβουμε κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα, οι ίδιοι οι νέοι θα διαρωτηθούν. Ωραία, αναλύετε το πρόβλημα και μιλάτε για το πρόβλημά μου, αλλά τι κάνετε για να το διορθώσετε. Και όταν είπα ότι η στρατηγική 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει και συγκυριακά μέτρα, αλλά και μακρόπνοα και διορατικά μέτρα, το θέμα της ε, απασχόλησης των νέων είναι θέμα άμεσο, βραχυπρόθεσμο και συγκυριακό. Και αν πιστεύουμε ότι οι μικροπιστώσεις μπορεί να είναι ένα καλό μήνυμα και μια καλή πολιτική για τους, ε, εργο... για τους επιχειρηματίες, θα μπορούσαμε το πρόγραμμα αυτό για τις μικροπιστώσεις να το κάνουμε πιο ελαστικό και να το εγκρίνουμε αν υπάρχει συνένεση, μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Επίσης υπάρχει θέμα και κατάρτισης, επιμόρφωσης και απασχόλησης. Αυτές οι πολιτικές θα προωθήσει η Ισπανική Προεδρία σε συνεργασία με τον νέο Επίτροπο για να δούμε τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να προτείνουμε για να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα η ανεργία επηρέασε πολύ πιο άμεσα και οδυνηρά τους μετανάστες και μάλιστα τους νέους μετανάστες. Αυτοί βιώνουν στο πετσί τους πολύ πιο έντονα το θέμα της ανεργίας. Οπότε σε ένα νέο μετανάστη πρέπει να δώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες ε, που έχει και ένας ε, άνεργος υπήκος του κράτους μέλους. Και εκεί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην επιμόρφωση, την κατάρτιση και την κοινωνική ένταξη. Δεν μπορεί να είναι περιθωριακό θέμα αυτό της ευκαιρίας προς τους νέους μετανάστες. Γιατί όντως αυτοί ε, έχουν ποσοστό ανεργίας πολύ ψηλότερο από τον ε, εθνικό μεσόρο. Η κυρία Χιμένες. Σε ό,τι αφορά τη φτώχεια, όντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι ένα λίκνο ευημερίας και ανάπτυξης, έχουμε παρόλα αυτά 80 εκατομμύρια φτωχούς και ομάδες κοινωνίας ε, ιδιαίτερα ευάλωτες. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη και την υποχρέωση να προωθήσουμε ενεργές κρατικές ή δημόσιες πολιτικές, ώστε σιγά σιγά να περιορίσουμε αυτού, στους θύλακες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Γνωρίζετε κυρίες και κύριοι ότι οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες. Παρ' όλα αυτά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούμε να συντονίσουμε τις πολιτικές μας. Και αυτός ο, αυτή η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού έχει αποφέρει καρπούς και ωφέλη σε τομείς. Για παράδειγμα, γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων και εκμετάλλευση των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να βελτιώσουμε τις προδιαγραφές κοινωνικής προστασίας αφενός και αφετέρου να συμπεριλάβουμε στο πολιτικό μας πρόγραμμα θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Όχι μόνο για να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση των προβλημάτων, αλλά και για να αυξήσουμε την ευαισθησία μας, την κοινωνική μας ευαισθησία, αλλά και την πολιτική μας ευαισθησία και να εγκύψουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και στις 21 του Ιανουαρίου που έγιναν τα εγγένεια αυτής της συνδιάσκεψης για την ανακήρυξη του 2010 ως έτους, Ευρωπαϊκού έτους ε, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο ίδιος ο πρόεδρος ε, της Ισπανικής κυβέρνησης, ο κ. Σαπατέρο, παρουσία του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μπαρόζο, εξέφρασε το μήνυμα όχι μόνο της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανάδειξης ε, αυτού του στόχου προτεραιότητα, αλλά είπε ότι στην ίδια τη στρατηγική του 2020 θα πρέπει ο στόχος να συμπεριληφθεί κοινωνική συνοχή και να είναι ακρογωνιαίος λίθος αυτού του νέου κοινωνικού και πολιτικού μοντέλου. Οπότε με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, που είναι βασική μέθοδος εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προωθήσουμε αυτό το θέμα και ταυτόχρονα ενεργές κρατικές πολιτικές, γιατί πολλές χώρες έχουν καταφέρει με τις πολιτικές τους να μειώσουν το χάσμα ε, μεταξύ των ε, φτωχών στρωμάτων της κοινωνίας. σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους με αναπηρίες, και εκεί σημειώθηκε πρόοδος τα τελευταία χρόνια και μάλιστα εντυπωσιακή. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν κρατικές πολιτικές που αποκατέστην την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών με αναπηρίες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δικό της επίπεδο κατάφερε να σημειώσει πρόοδο στα θέματα αυτά. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαράζει τη στρατηγική για την αναπηρία για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη έχουμε αρχίσει τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με το τρίο για να προωθήσουμε κάποιες πολιτικές απασχόλησεις. Το, κάνουμε, το εφαρμόζουμε ήδη στην Ισπανία και βλέπουμε ποιες πολιτικές χρειάζονται που θα μπορούσαν να γίνουν παράδειγμα εμείς και για τις άλλες χώρες, ώστε να προωθήσουμε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ανθρώπων με αναπηρίες. Θα διοργανώσουμε και μία υπουργική διάσκεψη στο Ισπανικό εξάμεινο και οι Υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας θα συνέλθουν για να ασχοληθούν με συγκεκριμένες πτυχές αυτής της στρατηγικής και με κάποια νέα στοιχεία που θα επεξεργαστούμε στις χώρες μας. Η διάσκεψη αυτή θα γίνει στις 19 Μαΐου στη Σαραγώσα. Επίσης θα συνεργαστούμε με όλες τις οργανώσεις και τα σωματεία αναπήρων. Γιατί αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή όλων αυτών των οργανώσεων. Έτσι θα ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, όπως μας ζητούν επίμονα αυτές οι οργανώσεις. Άλλωστε και η Βελγική Προεδρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα αυτά, ιδιαίτερα κατά πολέμηση της ένδυας. Θα καταλήξουμε λοιπόν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αποκινούμε τη Βελική και την Ουγγρική Προεδρία για θέματα κατά πολέμηση της φτώχειας και δικαιώματα των αναπήρων. Θέλουμε συγκεκριμένα εχέγγυα αλλά και αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Αΐντο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για το ενδιαφέρον που δείξατε για την ισότητα των φύλων και την ισότητα ευκαιριών. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ίση μεταχείριση, την καταπολέμηση τη διακριτική μεταχείριση, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση, από την πιο κατάφορη μέχρι την πιο εκλεπτισμένη, οφείλεται σε μία αδικία. Η αδικία είναι ασύμβατη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μία ένωση αξιών και ίσων δικαιωμάτων ε, των πολιτών τη. Γι' αυτό και είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στην πρόθεση αυτής της οδηγίας και σε ό,τι αφορά τις αναπηρίες. Πρέπει όλες οι χώρες να δείξουν συνέπεια σε ό,τι αφορά την προσχώρησή τους στην Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αναπήρων. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις υποδομές μας στα διάφορα κτίρια για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των αναπήρων και με αυτό το πνεύμα συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Φυσικά υπάρχουν επιφυλάξεις. Τώρα αρχίζουν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Ξεκίνησαν στις 22 Ιανουαρίου με την Ισπανική Προεδρία. Η επόμενη συνεδρία έχει προβλεφθεί για τα μέσα Φεβρουαρίου. Προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε κάπως τις ιδέες μας. Πάντως δυσκολίες υπάρχουν, δεν σας το κρύβω. Και το Συμβούλιο προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, γι' αυτό και δεν μπορώ να, να προεξοφλήσω την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Πάντως και εσείς μπορείτε στις χώρες σας να προωθήσετε τα πράγματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τη βία, την ερώτηση της κυρίας Λίν, σίγουρα υπάρχει βία στο σπίτι και προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Όχι μόνο στο σπίτι, γιατί η βία που ασκείται κατά των γυναικών μερικέ φορέ ασκείται ακριβώ επειδή είναι γυναίκε, λόγω του φίλου του. Και μάλιστα όχι μόνο εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέραν των συνόρων τη. Θα ασχοληθούμε με τη συναισθηματική βία, αλλά και με το σωματεμπόριο, με την ε, εκμετάλλευση των γυναικών για σεξουαλικούς ε, σκοπούς. Είναι μια νέα μορφή ε, σκλαβιάς και ξανδραποδισμού αυτή η μεταχείριση των γυναικών. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τέτοιες μορφές ε, σκλαβιάς, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον ε, γενετήσιο ακροτηριασμό. Είναι πολλές ε, οι μορφές βίας που ασκούνται κατά των γυναικών μόνο, μόνο εξαιτία του φίλου τους και αυτά είναι απαράδεκτα. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για, το, για τις μισθολογικές διαφορές, το μισθολογικό χάσμα, σίγουρα είναι μια ανυπόφορη μορφή διακριτικής μεταχείρισης, γι' αυτό και θα πρέπει να προωθήσουμε τη σταδιακή εξάλληψη αυτών των μισθολογικών διαφορών ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Βέβαια, δεν αρκούν οι νομοθετικές διατάξεις. Χρειαζόμαστε και ελεγκτικούς μηχανισμούς για να εξακριβώσουμε τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε στην Ισπανία τα Υπουργεία Εργασίας και Ισότητας ε, μέσω ενός πρωτοκόλλου με βάση το οποίο πραγματοποιήσαμε 5.000 ελέγχους στις ε, ισπανικές επιχειρήσεις για να εξακριβώσουμε την έλλειψη τέτοιου, τέτοιων μισθολογικών διαφορών. Χρειαζόμαστε λοιπόν και λογοδοσία και έλεγχο. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάποια φαλοκρατικά στερεότυπα στην παιδεία, στον ε, επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και στην άτυπη διάσκεψη υπουργών ισότητας που θα γίνει 25 και 26 Φεβρουαρίου στη Βαλένθια, η Ισπανική Προεδρία θα υποβάλει εν, μια προκαταρκτική έκθεση για τις μισθολογικές διαφορές που θα αποτελέσει βάση εργασίας και για τη Βελική Προεδρία που έχει αναγάγει αυτή τη μισθολογική διαφορά σε προτεραιότητα και την εξάλληψή της. Είναι σημαντική η συνεργασία των τριών προεδριών γιατί εξασφαλίζεται μια συνέχεια των ε, κοινοτικών προγραμμάτων για 18 μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τρίτη ομάδα ερωτήσεων και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρίσορτ Θαγκρού και μετά την κυρία Καρυμαντελή. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω θερμά τους Ισπανούς υπουργούς και Πιστεύω ότι και κατά το τέλος της Ισπανικής Προεδρίας θα είμαστε εξίσου ικανοποιημένοι όπως σήμερα, μετά τις εξαγγελίες για το Ισπανικό πρόγραμμα. Ήδη υπευλήθη μια πληθώρα ερωτήσεων προ του τρει υπουργού. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κορμπάτσο, που ήταν πολύ γενναιόδωρο για το χαρακτηρισμό τη συνθήκη τη Λισαβόνα ή τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Δεν θα ήθελα η στρατηγική του 2020 να γίνει μια αθολογία αγαθών προθέσεων όπω η στρατηγική τη Λισαβόνα. Γιατί η στρατηγική ε, της Λισαβόνας δεν ήταν ε, τραγωδία, ήταν τραγέλαφος. Πολλοί στόχοι, αλλά ελάχιστα επιτεύγματα. Θα προτιμούσε λοιπόν λιγότερη εξαγγελία προθέσεων και περισσότερα απτά αποτελέσματα. Αναφερθήκατε στα, στις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Μας κάνατε όμως μία παρουσίαση, σαν ήταν αυτή η οργάνωση ε, της παγκόσμια οργάνωση Εργασίας που ιδρύθηκε το 1919 σαν να είναι κάτι καινούριο, σαν να μην υπήρχε. Παράδειγμα, η οδηγία για το Ράριο εργασίας που ανέφερε ο Αλεχάνδρος Σέρκας. Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από το κάποιος αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οργάνωση της εργασίας, γιατί σχεδόν όλες οι χώρες μέλη κύρωσαν τις ε, συμβάσεις της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Και μία ερώτηση προς την Υπουργό που ονομάζεται Μπιμπιάνα. Αν θέλετε να γεφυρώσετε αυτό το μισθολογικό χάσμα, δεν θα ήταν καλύτερο να συστήσετε στα κράτη-μέλη να απαρνηθούν αυτή τη σύμβαση για το μισθό που είχε εγκριθεί πριν από άπειρα χρόνια, που ε, τότε μόνο οι, οι ε, εργάζονταν. Γιατί εκεί αναφέρεται ότι ο μισθός του άνδρα θα πρέπει να είναι ε, επαρκής ώστε να μπορεί να βιοπορίζεται από αυτό ολόκληρη η οικογένεια. Αυτή είναι μία από τις συμβάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να καταργηθεί. Να καταργηθεί και να μην λαμβάνεται πια υπόψη. Ευχαριστώ ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ε, να, να τροποποιηθεί λίγο λέγοντας ότι ο μισθός της γυναίκας ή του άνδρα θα καλύπτει τις ε, βιοποριστικές ανάγκες της οικογένειας. Κυρία Καρυμαντελή, καλημέρα και καλώς ορίσατε. Καλό κουράγιο πρώτα απ' όλα σας εύχομαι, γιατί έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι ε, η συμφιλίωση της Ευρώπης με τους ε, πολίτες. Ε, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων δεν ψήφισαν σε ευρωπαϊκές εκλογές γιατί δεν ανταποκρίνεται η Ευρώπη στις προσδοκίες τους και όσον αφορά τη στέγαση και όσον αφορά την εργασία και όσον αφορά ένα σωρό άλλα ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης. Λοιπόν, η στρατηγική της Λισαβόνας, το είπαν όλοι με κάθε τρόπο, ε, εστέφθη από αποτυχία. Η στρατηγική 2020 ε, παραμένει να δούμε τι θα κάνει. Κεντρικό ερώτημα που θέτω εγώ θα αναθεωρήσετε, θα αμφισβητήσετε αυτήν την έννοια αύξησης και ε, απόλυτα ε, μη επιτεύξιμης παραγωγικότητας που αναφέρονται εδώ και που προϋποθέτει εργαζόμενους που τους στίβουμε και τους πετάμε σαν λεμονόκουπες. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτησή μου. Δεύτερη ερώτηση η κοινωνική κρίση συμβαδίζει με την περιβαλλοντική κρίση. Σημαίνει αυτό ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές ε, εργασίας, αηφόρου, σταθερής και που δεν θα κλείνουν τα εργοστάσια για να πάνε κάπου αλλού, ε, σε κάποια άλλη περιοχή της γης, τότε θα πρέπει να ε, ε, επιλέξουμε την πράσινη οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη. Τι θα κάνετε σχετικά με αυτό. Αναφερθήκατε ε, στον στο έτος καταπολέμησης της ένδυας, πράγμα πολύ δύσκολο γιατί σύμφωνα με τη Λισαβόνα θα έπρεπε να είχε εκριζωθεί η ένδυα μέχρι το 2010. Επίσης, τι θα κάνετε όσον αφορά τη στέγη. Θα μιλήσετε ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ξέρουμε ότι η ενέργεια ε, ε, κοστίζει όλο και περισσότερο στους, στις οικογένειες. Και τέλος, θα προωθήσετε συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Ελιζαμπέτ Μογά και μετά ο κύριος Πουπάκης. Κυρία Μωρά, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτο ερώτημα σχετικά με την αναπηρία. Είπατε Ευτυχώς έχουμε δημόσιες πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε την αναπηρία. Όμως, κυρία Υπουργέ, βλέπουμε σήμερα ότι στις δημόσιες πολιτικές όντως ε, προβλέπονται κάποια ποσοστά για άτομα με αναπηρία, αλλά σπανίως εφαρμόζονται. Ερώτησης, τι θα κάνετε έτσι ώστε πρώτα απ' όλα οι δημόσιες πολιτικές να εφαρμόζονται όσον αφορά ε, τα άτομα με αναπηρία. Δεύτερη ερώτηση. Η καταπολέμηση της, ε, του αποκλεισμού, κυρίως δε του αποκλεισμού των νέων. Είπατε ότι είναι συγκυριακή η ενεργεία των νέων. Εγώ όμως δεν με την άποψή σας. Σήμερα είναι διαρθρωτική η ενεργεία των νέων και θα παραμείνει διαρθρωτική όσο επιτρέπουμε στους νέους να τελειώνουν την εκπαίδευσή τους χωρίς συγκεκριμένη κατάρτιση, χωρίς συγκεκριμένες δεξιότητες. Αυτή η κατάσταση θα τους αποκλείσει από την κοινωνία, θα τους αποκλείσει από την αγορά εργασίας τι προτίθεστε να κάνετε, τι σκέφτεστε ε, να κάνετε έτσι ώστε να ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα της έλλειψης κατάρτισης. Και να μην μου πείτε ότι το πρόβλημα αυτό είναι εθνικό ζήτημα. Όχι, είναι ευρωπαϊκό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν τέτοιο. Τελευταία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Ισότητα ανδρών γυναικών. Είπατε, κυρία Υπουργέ, ότι οι γυναίκες υπολείπονται όσον αφορά ε, το, τους μισθούς. Αλλά αυτή ε, η μισθολογική καθυστέρηση συνεπάγεται και καθυστέρηση στην καριέρα τους. Ε, και αυτό βεβαίως φαίνεται και στην σύνταξή τους τι θα κάνετε κύριε Υπουργέ έτσι ώστε να ξεπεραστεί αυτή η καθυστέρηση στις ε, καριέρες των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Πουπάκης και μετά είχα εγγράψει τον εαυτό μου αλλά νομίζω ότι θα παραχωρήσω τη θέση μου σε κάποιους άλλους. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λιζότο. Κύριος Πουπάκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους ε, κυρίους Υπουργούς για τη διάθεσή τους να μας ενημερώσουν. Ήθελα με δεδομένα τα υψηλά ποσοστά ανεργία στα κράτη-μέλη, την ανάγκη υιοθέτηση ενό νέου πλαισίου για την απασχόληση για να αποφύγουμε μια γενικευμένη κοινωνική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το απαιτούμενο για ενδυνάμωση τη κοινωνική προστασία με δημιουργία νέων και ποιοτικότερων θέσεων εργασία και την επανεξέταση τόσο των παθητικών όσο των ενεργητικών πολιτικών, να κάνω δύο ερωτήματα. Πρώτον, για τι προθέσει τη Ισπανική Προεδρία, για την αναγκαιότητα στήριξη των χαμηλών οικονομικά πληθυσμιακών στρωμάτων με ενίσχυση συγκεκριμένα των επιδομάτων ανεργίας και του πλέγματος της προνοιακής πολιτικής, όπως η βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και ένα δεύτερο ερώτημα, καθώς και τι είδους κατευθύνσεις για την υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, όπως ο επαγγελματικό προσανατολισμό, προγράμματα επανακατάρτιση, προγράμματα επαγγελματική κατάρτιση, σε αντικείμενα πάντα συμβατά με τι ανάγκε τη σημερινή ενόψη κρίση αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιζότο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και η Επιτροπή και ο Πρόεδρος Μπαρόζο ε, και ε, ο Επιτρόπος Αντόρα πολύ επιφανειακά ε, ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά που μας απασχολούν σήμερα. Και επίσης η Ισπανική κυβέρνηση ε, με πολύ σκληρό τρόπο αντιμετώπισε ε, την μετανάστευση και κυρίως την παράνομη μετανάστευση, αναφέρομαι στην απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2000. Ε, η Ισπανία, όπως και η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, έχετε ιδιαίτερα προβλήματα με την μετανάστευση. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήρθε η ώρα να ασχοληθεί η Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το θέμα αυτό και να μην το αφήσουμε στα χέρια των μεμονωμένων κρατών. Όσον αφορά τώρα την εργασία. ξέρετε ότι στην Ιταλία και νομίζω περισσότερο στην Ιταλία από ότι στην Ελλάδα ή στην Ισπανία οι πολίτες δεν δέχονται την απασχόληση των μεταναστών τη στιγμή που υπάρχουν άνεργοι ε, δικοί τους. Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Γιατί έχουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων πολιτών που είναι άνεργοι. Γιατί λοιπόν να ασχοληθούμε μόνο με τους άνεργους μετανάστες. Ε, Κύριε ε, Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ, πριν σας δώσω το λόγο, στις ε, ε, συνθήκες ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε είναι παρά να προχωρήσουμε με επικυρώσεις σε κάθε χώρα που μπορούν να οδηγήσουν σε ε, διαφορετική κατάσταση όσον αφορά τις επικυρώσεις. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσοι είχαν υπογράψει τις πρώτες συμβάσεις ε, να θεωρήσουμε ότι προχωρούν ε, κανονικά και με τις επόμενες. Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν έχετε ήδη κάποια απόφαση Τώρα, θέλετε μήπως να αλλάξουμε τη σειρά των απαντήσεων ή θέλετε να ε, απαντάτε πάντα γεωγραφικά όπως είσαστε καθισμένοι. Ό,τι θέλετε. Bueno, con a Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Φάλμπ μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα τεθεί αυτό το ζήτημα που θέσατε για τη ΔΟΕ, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Τώρα, οι μισθολογικές διαφορές είναι της τάξης του 17% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άλλωστε, η αναλογία των γυναικών στις ηθήνουσες θέσεις ή σε θέσεις λήψη αποφάσεων είναι μόνο 3%. Μια συμβολική ουσιαστικά παρουσία. Μόνο 3% των ε, εισηγμένων στη, στη στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις ε, έχουν ε, γυναίκες ε, διευθυντικά στελέχη ή μία στι δέκα γυναίκε είναι μόνο μέλη διοικητικών συμβουλίων σημαντικών επιχειρήσεων. Το 60% των αποφύτων πανεπιστημίων στην Ένωση είναι γυναίκε. και μάλιστα με πολύ καλύτερε επιδόσει από τους συμφοιτητές του άνδρες. Παρ' όλα αυτά έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση εργασία. Τα είπαμε όλα αυτά ε, ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελέσει εγκάρσια ε, προτεραιότητα της στρατηγικής του 2020 και όλων των φάσεων της απασχόλησης σε ό,τι αφορά την αναζήτηση, την προσπελασιμότητα, τη παραμονή στην αγορά εργασίας και φυσικά στην έξοδο από την αγορά εργασίας κατά τη ε, στιγμή της σύνταξης, κατά τη συνταξιοδότηση. Αυτά από μένα. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ο κύριος Κορμπάτσο. Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φάλμπρ. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σα. Πάντως, κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σα που είχατε την αυρότητα να την υποβάλλετε και στα ισπανικά. Θέσατε ένα ζήτημα ουσίας πραγματικά και ελπίζω και πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που προδιαγράψατε εσείς. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσει, να μην γίνει πραγματικά απλό ευχολόγιο η στρατηγική του 2020 και θα πρέπει, αν θέλουμε όλοι να έρθουν τα κοινωτικά θεσμικά όργανα κοντά στον πολίτη, να μην μένουμε οικειοθελώς απομακρυσμένοι από τα προβλήματά του και να χρησιμοποιούμε ορολογία που θα αγγίζει τον πολίτη. Θα πρέπει να περάσουμε από τις γενικότητες και τις αοριστολογίες σε συγκεκριμένα πράγματα θα πρέπει να συνεργαστούμε για όλα αυτά, γιατί είναι εύκολο να πετύχουμε συνένεση για τις γενικότητες. Αλλά η δυσκολία έγκυται μερικές φορές στην επίτευξη συγκεκριμένων λύσεων για τα ειδικά θέματα, όχι για τα γενικά και όριστα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει μεγαλύτερη ε, δυνατότητα αποφάσεων, περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες, περισσότερη συναπόφαση. Θα πρέπει λοιπόν όλοι από κοινού να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να μην είναι η νέα στρατηγική απλή συνέχεια της προηγούμενης. Δεν θέλω να επικρίνω κανένα, απλώς κάνω μια διαπίστωση. Η Ισπανική Προεδρία δεν είναι αφελής. Δεν μπορώ να σας α, υποσχεθώ ότι μέσα στο εξάμεινο θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι τουλάχιστον δύο θέματα θα συζητήσουμε στην Ευρώπη. Ένα θα είναι οι ιδέες και δεύτερο οι κατευθυντήριες γραμμέ και συγκεκριμένε οδηγίες. Και οι ιδέες και οι οδηγίες θα είναι σημαντικές, γιατί τώρα θα θέσουμε τα θεμέλια της Ευρώπης που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Και η Ισπανική Προεδρία είναι αποφασισμένη όχι απλώς να καταθέσει κάποιες ιδέες, αλλά να απηχήσει τις ιδέες των πολιτών και αυτές να καταθέσει στο τραπέζι. Το θέμα της ΔΟΕ, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η Ισπανική Προεδρία πιστεύει και ευελπιστώ ότι την άποψη αυτή θα την ασθενιστεί και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουμε ενεργά μέλη της ΔΟΕ. Και θα πρέπει σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα και τα οικονομικά και της απασχόλησης. Δεν μπορούμε να είμαστε απομονωμένοι, θα πρέπει να συμμετέχουμε σε μια παγκόσμια θεώρηση και να λαμβάνουμε υπόψη και τη ΔΟΕ. Τον Ιούλιο θα έχουμε την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και εκεί δεν θα παραστεί μόνο, αλλά θα έχει λόγο η Ισπανική Προεδρία. Και μάλιστα έχουμε μια κοινή διοργάνωση εκδήλωσης με τη ΔΟΕ, λίγο πριν την διάσκεψη των Υπουργών της G20 για την απασχόληση. Θα υπάρξουν λοιπόν πολλές επαφές και με τη ΔΟΕ. Στη δεύτερη σας ερώτηση, είπατε πώς θα συμφιλιώσουμε την Ευρώπη με τους πολίτες. Μα αυτή είναι η πραγματική πρόκληση. Θέλουμε να φέρουμε την Ευρώπη κοντά στους πολίτες. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές. Θα πρέπει το οικονομικό αυτό φρούριο που φτιάχνουμε στην Ευρώπη να μην καταστρέψει το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης. Γιατί στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπόδειγμα προς μίμηση. Όχι μόνο για τα οικονομικά θέματα, αλλά και για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αλλά και κυρίως για το κράτος πρόνοιας και την ευημερία της. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε όλοι, εξασφάλιση αυτού του μοντέλου. Σίγουρα οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να μην τις αγνοούμε. Μάλιστα, οι μελλοντικέ θέσει εργασίας θα πρέπει να σχετίζονται και με αυτό το θέμα. Θέλουμε πράσινες, φιλοπεριβαλλοντικές θέσεις απασχόλησης. Και δεν θα πρέπει αυτές να αγνοηθούν από τη στρατηγική του 2020. Τα προβλήματα της καταπολέμησης του αποκλεισμού δεν ξέρω αν παρερμηνεύτηκα, είπα ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια βραχυπρόθεσμα συγκυριακά μέτρα για να αποφευθεί η μετατροπή της ενεργείας των νέων σε διαρθρωτικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν επικεντρωθούμε μόνο στη συζήτηση της στρατηγικής για το 2020, για να χαράξουμε την Ευρώπη του 2020 και τη φανταστούμε και πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι η Ευρώπη του 2020, δεν θα πρέπει να αποσπαστούμε από το σήμερα, από την Ευρώπη του 2010, από την Ευρώπη του 2011, γιατί αν επικεντρωθούμε στα μακροπρόθεσμα και ξεχάσουμε τα βραχυπρόθεσμα, τότε είναι που θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες των πολιτών μας. Και το πρόβλημα των νέων είναι πραγματικά κέριο. Το θέμα της κατάρτισης, διατήρηση της επιμόρφωσης, απόκτηση δεξιοτήτων, αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, ένα νέο πλαίσιο για ποιοτική εργασία, ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών, αναφέρθηκαν τα επιδόματα. Θα προτιμούσα να μιλούμε για το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, που είναι αυτή η ευημερία. Ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας που σε περιόδους κρίσης θα πρέπει να εξαπλώνεται, να επεκτείνεται. Γιατί στους χαλεπούς καιρούς στην εποχή της κρίσης είναι που πλησιάζουν πολύ τα όρια της, ε, της φτώχειας και του αποκλεισμού και όχι σε περίπτωση παχιών αγελάδων. Στους δύσκολους καιρούς και στις αντίξωες συνθήκες χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη και αρρωγή οι πολίτες μας. Και τέλος, και σας ζητώ συγγνώμη πάλι πρόεδρε, γιατί μπορεί να μακρηγόρησα, το θέμα της μετανάστευσης θα πρέπει και αυτό να το εμβαθύνουμε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το αξιολογήσει, θα το επεξεργαστεί με τα κράτη-μέλη και τον Ιούνιο θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αντί να αναχαιτήσουμε τη μετανάστευση, καλύτερα να τη ρυθμίσουμε και να ευνοήσουμε την νόμιμη μετανάστευση. Γιατί η μετανάστευση σχετίζεται με την αγορά εργασία. και δεν θα πρέπει, και θα πρέπει η αγορά εργασίας να καθορίζει τις ανάγκες αυτής της ε, μετανάστευσης. Και αυτό θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη και νόμιμη, γιατί μια τέτοια μετανάστευση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη Ευρώπης και θα πρέπει ε, και οι μετανάστες να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων με τα αντίστοιχα των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο, τελευταία ομάδα εργασία. Α, η κυρία Χιμένε θέλει να πει κάτι συγγνώμη, γιατί μια ερώτηση είχε απευθυνθεί προς εμένα και θα ήθελα να την απαντήσω. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις απασχόλησης και τις θέσεις εργασίας γενικών για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Οι πολιτικές ε, για τους ανθρώπους με αναπηρίες είναι σημαντικές και έχουμε τρία επίπεδα. Έχουμε φυσικά το πρώτο επίπεδο που είναι το εθνικό και εκεί όλες οι χώρες θα πρέπει να έχουν ε, ενεργές, δραστήριες δημόσιες πολιτικές και να προβλέψουν κάποιες θέσεις για ανθρώπους με αναπηρίες. Και ήδη όλες οι χώρες έχουν κάποιες τέτοιες διατάξεις. Μπορεί να μην τηρούνται όλες. Πάντως καθημερινά υπάρχουν μεγαλύτερες, περισσότερες δεσμεύσεις και διαθεσιμότητα να αφιερωθούν ορισμένες θέσεις, να προβλεφθούν ορισμένες θέσεις για αναπήρωση. Και όλο και περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσει ε, προβλέπουν τέτοιε θέσει για ανθρώπου με αναπηρία. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πρόγραμμα φορολογικών ε, ναυσμάτων και κινήτρων που προώθησε ο Υπουργό Απασχόληση για τι επιχειρήσει που προσλαμβάνουν ανθρώπου με αναπηρίε. Υπάρχει βέβαια και το δεύτερο επίπεδο που είναι το ευρωπαϊκό. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, για του ανθρώπου με αναπηρία για την επόμενη δεκαετία. Και αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι δύο επόμενε προεδρίε, τη Βελγική και την Ουγγρική. Και στην Υπουργική Διάσκεψη τη Αραγώσα θα έχουμε συγκεκριμένε προτάσει. Α μην ξεχνούμε όμω τον ισχυρότερο μηχανισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα, που είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για του ανθρώπου με αναπηρίε. Αυτό ο μηχανισμό είναι πανίσχυρο. Τον έχουμε κυρώσει στην Ισπανία και πολλέ ε, χώρε μέλη έχουν κάνει το ίδιο. Και μάλιστα είναι υποχρεωτικό αυτός, αυτός ο μηχανισμός. Ανήκει πλέον στην Ισπανική Ένωμη και εκεί κατοχυρώνονται δικαιώματα για τους ανθρώπους με αναπηρίες και μάλιστα είναι υποχρεωτικής εφαρμογής και για να έχει κανείς πρόσβαση σε μια θέση απασχόλησης θα πρέπει να περάσει πρώτα τις πολιτικές επιμόρφωσης και κατάρτισης. Θα πρέπει και σε αυτό το θέμα να δώσουμε έμφαση και να συμπεριλάβουμε και τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Και για μια ερώτηση που απάντησε ο κύριο Κορμπάτζο, ο Υπουργός Κορμπάτζο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 2060, δηλαδή σε μια πεντηκονταετία, που μην, νομίζετε ότι είναι και πολύ μακριά, όταν θα σκεφτόμαστε τότε το μέλλον, θα έχουμε 152 εκατομμύρια ηλικιωμένου. άνω των 65 ετών. Χρειαζόμαστε λοιπόν εργατικό δυναμικό, χρειαζόμαστε μετανάστες, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί η Ευρώπη γερνάει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πλάμ και μετά η κυρία Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους τρεις υπουργούς που εκπροσωπούν την Ισπανική Προεδρία και να τους συγχαρώ για το πρόγραμμα το οποίο μας έχουν παρουσιάσει και που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, κυρίως όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Μας είπατε ότι θα πρέπει να καθορίσουμε το μέλλον το 2010, το 2011 και βεβαίως και το 2020. Νομίζω ότι οι στόχοι που προτείνεται για τα κοινωνικά ζητήματα, στόχοι προς την επίτευξη των οποίων ελπίζομαι ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεισφέρουμε αποτελεσματικά, ε, και ε, ε, χάρη στη στρατηγική την οποία ε, αυτή τη στιγμή εκπονούμε για το 2020, ελπίζουμε λέω ότι όλα αυτά θα έχουν θετική έκβαση. Θα ψηφίσουμε σύντομα για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση όσον αφορά την οδηγία για την, για την άδεια μητρότητος, για την οποία είμαι εγώ η συγγήτρια θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η προσέγγιση της Ισπανικής Προεδρίας όσον αφορά αυτήν την οδηγία. Την οδηγία δηλαδή που ασχολείται με την άδεια μητρότητος. Δεύτερη ερώτηση. Ο Πρωθυπουργό, ο κ. Θαπατέρο, αναφέρθηκε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σύμφωνο. Ποια είναι η προσέγγιση της Ισπανικής Προεδρίας όσον αφορά αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Ευχαριστώ πολύ πρέπει να πούμε ότι αναφέρεται η κυρία Πλάμ στις δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος ε, Θαπατέρο στην Ολομέλεια. Ναι, μια ερώτηση ε, που θίγει θέμα το οποίο ήδη έδεξαν πολλοί συνάδελφοι και επί του οποίου νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός από τις προτάσεις και της Ισπανικής Προεδρίας μεταξύ άλλων. Με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα ε, την δέσμευση της Ισπανικής Προεδρίας διαστόματος των Υπουργών. Αναφέρομαι στην ανεργία των νέων αλλά και στο δυναμικό των νέων. Νομίζω ότι ορθώς πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα των νέων και της ενεργείας των νέων δεν είναι πλέον συγκυριακό, είναι εγκάρσιο και είναι και διαρθρωτικό. Ε, και ε, νομίζω ότι αφορά νέους ε, κάθε κοινωνικής προέλευσης. Δεν είναι καθόλου συγκυριακό. Πιστεύω λοιπόν ότι και όσον αφορά τον συντονισμό αλλά και όσον αφορά μελλοντικές οδηγίες για την απασχόληση θα πρέπει να δούμε το εγκάρσιο του ζητήματος. Ας πούμε, όσον αφορά το, τα προνοιακά συστήματα. Θα πρέπει οι νέοι να έχουν κυρίαρχη θέση ε, και όπως είπε και ο υπουργό, θα πρέπει να προβληθεί ένα δίκτυο προστασίας το οποίο θα ακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι την, το τέλος της ζωής του. Της ζωής του. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα ε, να μην προβλεφθούν επιδόματα, ε, δηλαδή ε, μπορούν, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Αντιθέτως πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ακόμα και σε επιχειρήσεις για τους νέους. Κίνητρα επίσης για την στέγαση ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ναι τα προβλήματα τα οποία είναι συγκυριακά και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη αλλά όμως ταυτόχρονα να ληφθούν και ε, ε, μέρημνες για την τελική λύση του προβλήματος. Πρόεδρος, δύο ερωτήσεις. Πρώτον για τη στρατηγική 2020. Το ακούσατε ότι υπάρχει μία δυσφορία στα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η στρατηγική 2020 και σχετικά με τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην συζήτηση. Βεβαίως γνωρίζομαι ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων δεν έχει ακόμα οριστεί και επομένως δεν έχει ακόμα σκύψει πάνω στο θέμα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά την απασχόληση. Et notamment σε όλα τα τμήματα της αγοράς εργασίας ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία πρόσβασης των νέων. Δύσκολα οι νέοι μπαίνουν στην ε, αγορά εργασίας. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι στην ηλικία των 50-55 ετών χάνουν την εργασία τους. Απ' την άλλη πλευρά γνωρίζομαι ότι η προοπτική ανάπτυξης ε, δεν θα ξεπεράσει το 2%, άρα η δυσκολία δημιουργίας θέσεων εργασίας ε, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Επομένως, ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα το θέμα της απασχόλησης στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και όχι, ένα, και όχι μία παρεμπίπτουσα πολιτική των λοιπών πολιτικών ε, ή ας πούμε ε, σκεπτόμενοι ότι η ανάπτυξη θα δώσει αυτόματα λύσεις στο θέμα της ε, απασχόλησης. Επίσης, ένα τρίτο ζήτημα γνωρίζετε ότι η αναπτυξη θα δωσει αυτοματα λύση στο θεμα της Λισαβόνας εισήγαγε μια νέα νομική βάση όσον αφορά την δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από τη μία χώρα της Ευρώπης στην άλλη. Η Ισπανική Προεδρία θα ε, ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξανανοίξει η συζήτηση έτσι ώστε μια σωστή νομική βάση να εξευρεθεί όσο γίνεται γρηγορότερα. Θα σας δώσω το λόγο για το τελευταίο τμήμα, ε, το τελευταίο ομάδα ερωτήσεων. Πρεσιδέντα... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Bien, la primera pregunta. και μία ερώτηση. που αποτελούνταν από τα δύο τμήματα. Το πρώτο θα το απαντήσει η συνάδελφος Χιμένες. Το δεύτερο αφορούσε το κοινωνικό σύμφωνο. Είναι δική μου αρμοδιότητα και αναφέρθηκε και στην ε, ανακτήρια ομιλία του Πρόεδρου Σαπατέρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα αύριο το πρωί θα συνεδριάσει στη Βαρκελόνη η Κοινωνική Τρόικα. Και σήμερα το απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνάντηση της Κοινωνικής Τρόικας στη Βαρκελόνη. Αύριο θα διεξαχθεί η άτυπη συνεδρίαση της Τρόικας. Και μάλιστα η Προεδρία ήδη είχε διαβουλεύσει με τους κοινωνικούς εταίρους. Και εξετάζουμε την ιδέα ενός κοινωνικού συμφώνου, γιατί η οικονομική κρίση και η κρίση της απασχόλησης θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ε, συμμετοχής και της ανάμειξης των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών και των εργαζομένων. Το θέμα του τεράστιου δυναμικού των νέων και το πρόβλημα της ανεργίας των νέων που είναι εγκάρσιο. Συμφωνώ απόλυτα. Όντως, είναι καθολικό αυτό το πρόβλημα και φυσικά δεν είναι μόνο οι νέοι που έχουν πληγεί από την ανεργία, αλλά σίγουρα όταν είναι κανείς νέος και ανειδίκευτος επιπλέον, τότε είναι που η ανεργία είναι πολύ πιο υψηλή. Οι μελλοντικέ δε του νέου αυτού είναι πολύ μικρές. Γι' αυτό και η απάντηση δεν θα πρέπει να είναι μόνο σε επίπεδο απασχόληση, αλλά και σε νωρίτερη φάση τη επιμόρφωση και τη κατάρτιση, για να αποκτήσει ο νέο δεξιότητε και προσόντα. Όταν ένα νέο ε, δεν ολοκλήρωσε τις σπουδέ του ή τις εγκατέλειψε, θα πρέπει στις προσπάθειες επασχόλησης να προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε το ενδιαφέρον του νέου, να επιστρέψει και στις σπουδέ, να συνεχίσει την επιμόρφωση και την κατάρτισή του. Θα πρέπει να δοθούν ενάψματα προς τους νέους και σε επίπεδο κατάρτισης και επιμόρφωσης και μετά σε επίπεδο απασχόλησης. Οποιοδήποτε μέτρο που θα εξάψει την περιέργεια των νέων και θα το επαναφέρει στα θρανία ώστε να συνεχίσει την κατάρτισή του είναι θετικό. Η πρόεδρος μίλησε για τις δυσκολίες πρόσβασης ε, που έχουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Συμφωνώ μαζί σας κυρία Πρόεδρε, πάντως είναι προφανές ότι η στρατηγική 2020 ε, δεν μπορεί να ξεχνά την οικονομική κρίση. Πότε ε, θα ξεφύγουμε από την κρίση, όταν θα έχουμε εξομαλύνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα ή όταν θα μπορέσει η νέα οικονομία να ανακτήσει τις θέσεις απασχόλησης που κατήργησε η κρίση. Αυτό είναι σημαντικό θέμα, γιατί η κρίση κατά τη γνώμη μας δεν θα ξεπεραστεί όσο δεν έχουμε επαναφέρει στην αγορά εργασίας όλα τα εκατομμύρια των ανέργων που έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της κρίσης. Βέβαια, ίσως υπάρξει ο πειρασμός να θεωρήσουμε ως λήξασα την κρίση ε, όταν ανακάμψουν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, όταν θεωρήσουμε ότι η οικονομική κρίση έχει ξεπεραστεί επειδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ξαναστάθηκαν στα πόδια τους. Αλλά αν μιλούμε για στρατηγική της Λισαβόνας και ξεχνούμε την ε, στρατηγική της απασχόλησης ως προτεραιότητα, είναι ε, σαν να μιλάμε κινέζικα και κανένας πολίτης δεν θα μας καταλάβει. Αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη, κυρία Πρόεδρε. Όταν χαράξουμε τη στρατηγική του 2020, θα πρέπει να δώσουμε απτές απαντήσεις στα προβλήματα που μαστίζουν τον Ευρωπαίο πολίτη. Και το φλέγον ζήτημα σήμερα για τον πολίτη είναι η απασχόληση, είναι η ανεργία. Η ανεργία ή ο φόβος της απώλειας της θέσης απασχόλησης. Αυτά τα απτά ζητήματα θα πρέπει να θέσει ως επίκεντρο η στρατηγική του 2020. Και το θέμα των συντάξεων επίσης. Φυσικά είμαστε πρόθυμοι για συνεργασία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την ανέβρεση μιας νέας μετά την ε, διαμόρφωση των νέων νομικών βάσεων. κυρία Αΐντο, σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω στην ερώτηση για την οδηγία της μητρότητας. Η Ισπανική Προεδρία εστερνίζεται πλήρως ε, την πρόταση για την προστασία της υγείας ε, των ε, γυναικών, εγγύων, λεχώνων και γαλοχουσών. Θα προωθήσουμε την οδηγία αυτή αναζητώντα ισορροπία μεταξύ διαφόρων πτυχών. η διάρκεια τη άδεια μητρότητα, η αμοιβή, οι αποδοχέ τη άδεια, η ένταση τη άδεια, η εξασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων των γυναικών μεταξύ της, της ε, γημοσύνης ε, του τοκετού και της ε, έναρξης της άδειας μητρότητας, η στιγμή της έναρξης άδειας μητρότητας, όλα αυτά είναι ε, θέματα που θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Θα πρέπει, έχοντας υπόψη τη συνυπευθυνότητα, να εξετάσουμε όλα αυτά τα συστήματα. Η οδηγία για την άδεια μητρότητας είναι προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας. Θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη ξεκινήσει τις δραστηριότητες αλλά από σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένουμε τις γνωμοδοτήσει και τη σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως την έκθεση της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων τη Γυναίκας τη 25 η Φεβρουαρίου. Θα περιμένουμε λοιπόν την έκθεση και τις γνωμοδοτήσει του Συμβουλίου και θα έχουμε στενή συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μαζί σα, ευελπιστώντα ότι θα καταφέρουμε να εναρμονίσουμε το επίπεδο προστασία. Ε, των εγγύων λεχόνων και γαλουχουσών γυναικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ε, Κύριε Υπουργή, θερμά σας ευχαριστώ και κυρίε Υπουργή, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είδατε το ζωηρό ενδιαφέρον των Ευρωβουλευτών και νομίζω ότι αυτό το ενδιαφέρον ε, ανταποκρίνεται στις τεράστιες προσδοκίες και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για τα κοινωνικά ζητήματα, ειδικά μετά την κρίση. Αύριο θα γίνει το άτυπο Συμβούλιο της Βαρκελόνης. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία σας και στο εξαμεινό σας και σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Chers collègues, je vous demande de reprendre place. Καθίστε παρακαλώ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Et ouvrir notre séance de vote. Je vous Ξεκινούμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες θα πρέπει να έχετε τις ε, κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι τις ξέχασαν και θέλουν τώρα να μας το πούν. Για κοιτάξτε, έχετε τις κάρτες σας όλοι. Tout est Όλα καλά, λέει η πρόεδρος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε άψογα. Επομένως, σημείο 14 της ημερησίας διατάξεως. Ψηφοφορία επί της ε, γνωμοδότησης της κυρίας Ροβάνα Πλάμ που τροποποιεί την ε, οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας για την εργασία των εγγύων λεχώνων και γαλγουσών εργαζομένων. Τροπολογία Κορνέλη είναι Πριν αρχίσουμε θα... Ε, ένα διαδικαστικό. Ποιο είναι το πρόβλημα, κυρία Κορνέλισεν. Όπως σας είπα χτες, ήταν πολύ συνήθιστη διαδικασία για τις ε, συμβιβαστικέ τροπολογίες και θα ήθελα ορισμένε διευκρινήσεις ε, για τους συμβιβασμούς. Η συζήτηση έχει κλείσει, λέει η και δεν θα ξαναρχίσουμε. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 48 υπέρ. Ε, ε, είναι διαδικαστικό. Όχι, λέει η Πρόεδρος, δεν φαίνεται καθόλου να είναι διαδικαστικό. Έχετε κάποιο κανονικό διαδικαστικό. Um, compromise A and B. Συμβιβασμός Α και Β έχουν γίνει από το συγητή με δύο ευρωβουλευτές που δεν έχουν υποβάλει τροπολογίες, κυρία Κονή και η κυρία Χίρς. Αυτοί δεν είναι, δεν είναι κανονικές συμβιβαστικές τροπολογίες και δεν θα πρέπει να χαρακτοριστούν έτσι. Και οι συμβιβαστικές D και F είναι τροπολογίες, όχι συμβιβαστικέ. Εντάξει, καταγράψαμε την αντίδρασή σας και ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εψήφισε ένας παραπάνω. Τώρα θα τα δούμε όλα στο μηχάνημα. Θα μας πει ποιος είναι αυτό. Α, τώρα εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει, πέρα της ψηφοφορίας. 23 ψήφοι υπέρ 25 κατά, επομένως απορρίπτεται η τροπολογία. Χωρί μικρόφωνο η πρόεδρο. δεν την ακούν οι διερμηνεί. εξακολουθεί χωρί μικρόφωνο. Λοιπόν, να παρακαλέσω ε, να ελέγξετε ότι κάθε ομάδα έχει του ψηφοφόρου που πρέπει. Τροπολογία 62 τη κυρία Ροντζόλη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 Ροντζούλη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 της κυρίας Πλάμ υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν όλοι υπάρχει ένας επιπλέον από το ΕΛΚ ένας ε, τελευταίος ένα μέλος αναπληρωματικό από το ΕΛΚ. Εψήφισε ένα από το ΕΛΚ παραπάνω, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη. Εγώ αντικαθιστώ την κυρία Ζωβιέσκα, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα μπορώ να μην ψηφίζω. Monsieur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 Ναι, αλλά πρέπει κάθε φορά να μου λέτε αν ψηφίζετε υπέρ, κατά ή αποχή. Euh, Ωραία, λύσαμε το ζήτημα τη της ε, ψήφου του ΕΛΚΑ. Επομένως, πέρασε. τη ψηφοφορία της ψηφοφορίας και παρακαλώ να μου πείτε με ποιο τρόπο ψηφίζετε, κύριε Σιμάσκη. Υπέρ. Ωραία. Πέρασε της ψηφοφορίας 23 υπέρ 25 κατά. Επομένως η τροπολογία αυτή δεν γίνεται δεκτή. Τροπολογία 13 και 44 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 1466 ταυτόσημα υπέρ κατά αποχές Επομένως εγκρίνεται η τροπολογία 65 καταπίπτει και φτάνουμε στις τροπολογίες 15 και 67 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 16 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. τροπολογία 17 έχει αποσυρθεί. τροπολογία 28 της εισηγητρίας υπέρ. Θέλετε επαλήθευση? Τι θέλετε να επαληθεύσετε λέει η πρόεδρος. Ωραία. Επί του τροπολογία 16 άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 16, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρασες της ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ. Α, εσείς ψηφίζετε υπέρ. Επομένως, 29 ε, ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Έχετε δίκιο. Εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. Η τροπολογία 17 απεσύρθη. Η τροπολογία 68 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 απεσύρθη. Τροπολογία 69 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πώς ψηφίζετε εσείς κύριε Σιμάσκη. Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 21 ψηφί κατά, εγκρίνεται. Τροπολογίες 19 και 20 αποσύρθηκαν. Τροπολογία 70 της Σίτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, τώρα έχει την ε, κάρτα του. Πάρα πολύ ωραία. Πέρα της πληροφορίες. 23 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, επομένως η τροπολογία 70 απορρίπτεται. Τροπολογία 21 απεσύρθη, τροπολογία 71 της ΣΥΤΡΙΑΣ υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Στροπολογία 72 της συγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 της συγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 της συγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 Ωραία, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 22, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 23 ε, υπέρ, 25 κατά. Έχετε δίκιο, απορρίπτεται. Τροπολογία 22 της συγγετρίας υπέρ. Κατά. Αποχέσε. Θέλετε να γίνει η επαλήθευση, νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. ψήφι κατά 26, ε, ε, συγγνώμη, υπέρ, 26 κατά, όντως απερίφθη. Τροπολογία 74, Ροντζόλη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 75 ε, της συγγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 76 της συγγητρίας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 77 της συζήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 79 ε, της υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 24 έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία 80 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 81 της κυρίας Κορνέλησεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 82 Τόμας Μάν υπέρ. Κατά. Το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 82 Τόμας Μάν. Εψήφισαν όλοι πέρα της 26 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Επομένως, η τροπολογία 82 εγκρίνεται. Τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής και ψηφίζουμε ένα πρώτο, μια πρώτη συμβιβαστική ε, τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται το α. Τροπολογία 25 Τόμας Μαν. Επ' αυτού υπάρχει αίτημα για χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 85 από το With Respect μέχρι την οδηγία 96-34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα από The Remuneration for μέχρι Calculated υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε την τροπολογία 26 του κυρίου Μάρτιν Κάστλερ υπέρ, κατά, αποχές, επίσης απορρίπτεται. Φτάνουμε τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία Β από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 96 της κυρίας Ροντζόλη υπέρ κατά αποχές η τροπολογία 96 της κυρίας Ροντζόλη δεν απεσύρθη. μονάχα η τροπολογία 28 της κυρίας Πλάμα απεσύρθη. Επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 96 της κυρίας Ροντζόλη. Μήπως οι επικεφαλείς ε, των ομάδων να ε, ε, δείχνουν την ψήφο. Όχι, όχι, λέει κύριε Ροτζολικό, είχα αποσύρει, είχα αποσύρει την τροπολογία μου. Αυτό ήταν καλά φυλαγμένο μυστικό του ΕΛΚ. Λοιπόν, τροπολογία ΟΜΕΝ ΡΟΙΤΕΝ υπέρ κατά εγκρίνεται. Αποχές, λέει η Πρόεδρος, το ξέχασα. Τροπολογία 95 της κυρίας Ραπτή και της κυρίας Παλιαδέλη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 98 ομιν Ρόιτεν, υπέρ, κατά, Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά, επομένως συγκρίνεται. Τροπολογία 99, Νάντζα Χίρς, υπέρ. Κατά. αποχέσε Απορρίπτεται σαφώς. Συμβιβασμό γάμα. Από τέσσερις ομάδες, αν και δεν είναι πολύ σαφές, υπέρ. Κατά. αποχέσε εγκρίνεται. Επομένως, τροπολογία διαγραφής 103 και 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές Τροπολογία 31, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 105 του κύριου Τόμας Μαν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 Τόμας Μαν και Κάσλερ υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. 25 υπέρ, 23 κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 33 της 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Πολύ ωραία. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. 25 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 109 του κυρίου Τόμας Μαν υπέρ Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρο. Γύρισα πολύ γρήγορα τη σελίδα μου. Τροπολογία 107 τη κυρία Κορνέλισεν. Ε, κατά δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το σύνολο χωρίς τη λέξη compulsory υποχρεωτικά υπέρ κατά. Αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. πέρας της ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, επομένως απορρίπτεται. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 108 της κυρίας Φιγκερέιδο. Θα ψηφίσουμε «Χωρίς of which two shall be obligatory», εκ των οποίων οι δύο θα είναι υποχρεωτικές. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές. Νομίζω πως είναι το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 23 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, επομένως απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει, επομένως. Φτάνουμε στην τροπολογία 109 του κυρίου Τόμας Μάν, τροπολογία διαγραφής υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 109, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο λοιπόν του άρθρου 10 και το ψηφίζουμε σε τέσσερα τμήματα. Σε τέσσερα τμήματα λοιπόν. Θα ψηφίσουμε πρώτα την εισαγωγή και την παράγραφο 1 υπέρ. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 10. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία σύγχυση. Ψηφίσαμε την κατάργηση του άρθρου 10. Οπότε, γιατί να ψηφίσουμε πάλι. Εκτός και αν έκανα λάθος για το νόημα της ψηφοφορίας. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Με, κυρία Φιγερέδο, να σας πω απορρίψαμε την τροπολογία του κυρίου Τόμας Μαν που, ήταν, ε, ε, που ήθελε διαγραφή του άρθρου 10. Όμως, επί του αρχικού κειμένου της ε, Επιτροπής έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία, ψηφοφορία κατά τμήματα. Και επομένως ψηφίζουμε τώρα επί του αρχικού κειμένου του άρθρου 10, έτσι όπως προκύπτει από την πρόταση της Κομισιόν. so Καλώς ε, το διευκρινίσαμε. Οπότε τώρα θα ψηφίσουμε αν συμφωνούμε με κάθε επιμέρους παράγραφο του άρθρου αυτού. Έτσι. Δεν ψηφίζουμε τη διαγραφή, ψηφίζουμε την αρχική παράγραφο. Θα ψηφίσουμε την κάθε παράγραφο χωριστά. Εγώ το αντίθετο είχα καταλάβει. Ότι θα ψηφίσαμε τη διαγραφή του κάθε σημείου. Όχι. Δεν θα ψηφίσουμε τη διαγραφή, θα ψηφίσουμε κάθε παράγραφο. Καλό θα είναι για να διευκρινίσουμε την ψηφοφορία. Ναι, ναι. θα τοποθετηθούμε επί κάθε παραγράφου υπέρ ή κατά. Νομίζω πως τώρα είναι σαφές. Θέλετε όμως περαιτέρω αποσαφήνιση, κυρία η συγκήτρια. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να αποσαφηνίσω την κατάσταση για την τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Τόμας Μάν, η ομάδα Άλτε ζήτησε χωριστή ψηφοφορία. Ψηφοφορία κατά τμήματα και μάλιστα σε τέσσερα τμήματα. Επομένως, από τη στιγμή από τη στιγμή που απορρίψαμε την απόρριψη, άρα έχουμε απορρίψει και κάθε τμήμα. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, λέει η πρόεδρος. Η τροπολογία του κυρίου Μαν αποσκοπούσε σε πλήρη διαγραφή του άρθρου 10. Εάν είχαμε υπερψηφίσει λοιπόν την τροπολογία του κυρίου Μαν, δεν θα υπήρχε πλέον άρθρο 10. Όμως εξακολουθεί και υπάρχει το άρθρο 10. Και επί του άρθρου 10 και επί του αρχικού κειμένου του άρθρου 10, η ομάδα Άλντε μας ζήτησε χωριστή ψηφοφορία, άρα ψηφίζουμε. Επομένως, εισαγωγή και πρώτο, ε, πρώτη παράγραφος ε, του αρχικού κειμένου της Κομισιόν του άρθρου 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Δεύτερη παράγραφος υπέρ. Κατά. Αποχές, το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, the member make points 1 and 2. Υπέρ κατά αποχές το τρίτο τμήμα εγκρίνεται το υπόλοιπο του κειμένου υπέρ κατά αποχές. Επίσης εγκρίνεται πάρα πολύ ωραία, επομένως το άρθρο 10 του αρχικού κειμένου του εγγράφου της Επιτροπής γίνεται δεκτό, ακέραιο και χωρίς καμία τροποποίηση. Τροπολογία 110 της κυρίας Φιγκερέδο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. Τροπολογία 114. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μυστικό καλά φυλαγμένο. Και αυτή την τροπολογία την έχω αποσύρει. Εγώ είχα στείλει τη σχετική ειδοποίηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λέτε γιατί δεν θα τα ψηφίσουμε λοιπόν. 114 ε, και 111 έχουν αποσυρθεί. Τροπολογία 113 της κυρίας Όμεν Ρόιτεν υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 21 ψήφοι υπέρ 26 κατά, επομένως η τροπολογία 113 δεν εγκρίνεται. τροπολογία 112 Μάρτιν Κάσλερ υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 115 Κορνέλισεν υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35 της συζητρίας υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 της ηγετρίας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 116 Τόμας Μαν υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι, μάλλον να μην πω ότι νομίζω, να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση λέει η Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 24 υπέρ 23 κατά. Εγκρίνεται. Ε δεν μπορούσε να είναι και σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 117 της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές ε, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 24 ε, κατά και επομένως η τροπολογία 117 απορρίπτεται. 118 της εισηγητρίας. Κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες 29 υπέρ 19 κατά. Επομένως η τροπολογία αυτή σαφώς εγκρίνεται. Τροπολογία 119 Μάρτιν Κάσλερ υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. 25 υπέρ 22 κατά, επομένως εγκρίνεται τροπολογία 120 της ε, εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική λύση δέλτα ε, και εδώ αναφέρεται μονάχα η εισηγήτρια ως ε, συγγραφέα αλλά υπέρ κατά αποχές ε, το ΔΕΛΤΑ εγκρίνεται. Τροπολογία 38 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 122 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123 Τόμας Μάν αυτό καταπίπτει. Το ίδιο και η τροπολογία 124. Ψηφίζουμε την 125 της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 41 της εισηγητρίας με μια προφορική τροπολογία η οποία θέλει να διαγράψει το σύζυγος ή ε, και τη σύντροφος κτλ. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 21 ψήφι περί 27 κατά, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 41 42 της ε, συγκεκρίας ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 Κρίστενσεν υπέρ. Α, αυτό είναι ένα άλλο μυστικό των σοσιαλιστών. Ψηφίζουμε λοιπόν στις τροπολογίες 128, 129, 130 υπέρ κατά. Θα επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 22 κατά, επομένως οι τροπολογίες 128, 129, 130 που είναι τροπολογίες διαγραφής εγκρίνονται επομένως το, άρθρο 12α καταπίπτει. Τροπολογία 131 της κυρίας Όμιν Ρόιτεν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 132 του κυρίου Πουπάκη, ε, τροπολογία διαγραφής υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Νομίζω ότι είναι σαφές το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, ε, τροπολογία 133 της, των κυριών Ράπτικ Παγαλιαδέλη υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται επίσης τροπολογία 43 της κυρίας Πλάμ υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Τροπολογία 43 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι υπέρ της ψηφοφορία. 25 υπέρ, 23 κατά, επομένω εγκρίνεται. Τροπολογία 134 του κυρίου Πουπάκη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 135 του ιδίου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 136 των κυρίων Τόμας Μάν και Μάρτιν Κάσλερ, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 136. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 25 υπέρ 23 κατά, επομένως τροπολογία 136 εγκρίνεται με δύο, με δύο ψήφους διαφορά που βλέπουμε συχνά στο αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορία. 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 44 της εισηγητρίας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εντάξει, επαλήθευση επί της τροπολογίας 44, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρασε. Η 21 ψήφοι υπέρ 27 κατά. Ε, έχετε δίκιο. Όχι, διορθώνει η Έχω εγώ δίκιο. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47 της συγκεκριτρίας γιατί 45-46 έχουν αποσυρθεί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία λοιπόν, ε, τροπολογία λέγω 49 η οποία διορθώθηκε έτσι ώστε να γίνει συνεκτική με το υπόλοιπο κείμενο. Τροπολογία 49, ούτως τροποποιηθήσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 του κυρίου Τόμας Μάν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 της συγητρίας υπέρ κατά αποχές νομίζω πως έχει αποσυρθεί αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Τροπολογία 2 λοιπόν ψηφίζουμε. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Επομένως η τροπολογία 2 εγκρίνεται. τροπολογία 59 Τόμας Μάν υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 51. Ψήφισαν όλοι υπέρα τη ψηφοφορία. 22 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, επομένω απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της συγγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 του κυρίου Τόμας Μάν υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 4 της συγγητρίας υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε λοιπόν επί της τροπολογίας 4 άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρασε. 24 ψήφοι υπέρ, 24 ψήφοι κατά. Πολύ καλά κάναμε και ε, επαληθεύσαμε, δεν εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 έχει αποσυρθεί, η τροπολογία 53 της κοινίας Νάτζα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 54 απεσύρθη, η τροπολογία 55 το Mann υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 το Mann υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της συγητρίας υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Τροπολογία 6, λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, 23 ψήφοι κατά, ω ε, συνήθω με δύο ψήφους διαφορά εγκρίνεται. Φτάνουμε στην τροπολογία 7 της συγγετρίας, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 πάλι τη ηγετρία υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ε, ή... Α, θέλετε επαλήθευση από του 57. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας. 25 υπέρ, 23 κατά, έχετε δίκιο, εγκρίνεται. Δεν ήταν σαφές όμως. Ε, λοιπόν, συμβιβασμός ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 της κυρίας Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 της ηγετρίας ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές η εισηγήτρια λέει ότι εγκρίνεται, αλλά μήπως να κάνουμε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας κάνουμε μια επαλήθευση παρόλα αυτά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, εδώ ξαφνικά έγινε πάρα πολύ σαφές το αποτέλεσμα. 42 ψήφοι υπέρ, ε, πέντε ψήφοι κατά, σαφέστατα εγκρίνεται. Ε, λοιπόν, τώρα ε, έχω εδώ μία πάρα πολύ περίεργη συμβαστική F, η οποία αναφέρεται μονάχα με έναν άνθρωπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 της συγκεντρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε το σύνολο τη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας ε, κυρία Ούμεν Ρόιτερ, αν βγάλετε την κάρτα σας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφοφορίας, δεν θα καταγραφεί η ψήφο σας. 31 ψήφοι υπέρ, 11 κατά 5 αποχές. Επομένως, η γνωμοδότηση της κυρίας Πλάμα εγκρίνεται και νομίζω ότι μπορούμε να τη συγχαρούμε. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Και περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία μας. Την πρόταση ψηφίσματος της κυρίας Λίνα. Παρακαλώ όσοι θέλουν να φύγουν από την αίθουσα να το κάνουν χωρίς πολύ φασαρία. Παράγραφος 2α9, τροπολογία 4 της κυρίας του κυρίου μάλλον, ε, συγγνώμη λέει πρόεδρος, του κυρίου Μπαλντασάρ. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πέντε. Ποιος είναι υπέρ του ίδιου, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ ιδιωτικέ συνομιλίε εκτό τη αίθουσα. Τροπολογία 6, Στέφαν Χιού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία Μπαλτασάρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Για τι αιτιολογικέ σκέψεις, πρώτη συμβαστική τροπολογία 2. Συντακτών Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχε. εγκρίνεται. Δεύτερη συμβαστική τροπολογία των ιδίων. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του κυρίου Μπαλτασάρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Ε, γιατί να κάνουμε ηλεκτρονικό ψήφο. Εδώ βλέπω ομοφωνία σχεδόν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται με μία αποχή μόνο το ψήφισμα της κυρίας Λίν. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Λίν. Nous en venons à notre dernier Και τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα το πρωί αφορά την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Για μια συγκεκριμένη περίπτωση της αιτήσει της Γερμανίας και της Λιθουανίας για τις επιχειρήσεις Κάρμαν και Σνέιτζ. Ποιος είναι υπέρ των δύο των επιστολών. Κατά αποχές, οπότε οι επιστολές θα διαβαστούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Διεκπαιρεώσαμε τις ψηφοφορίες μας και σας προτείνω να περάσουμε στα σημεία 17 και 18 για κοινή συζήτηση των δύο σημείων όπως είχαμε συμφωνήσει. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο για το σημείο 17 το συντάκτη της γνωμοδοτησής μας, τον κύριο Όλε Κρίστενσεν. Θα μας ενημερώσει για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, καθώς και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Thank you very much, Chairman. Excessive. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε η ακραία ανάληψη... Ε, Συγγνώμη κύριε Σιγητά, κανείς δεν σας ακούει αυτή τη στιγμή. Θέρμο παρακαλώ, τα πηγαδάκια και ιδιωτικέ συνομιλίε εκτός της αιθούσης, παρακαλώ. Λίγη ησυχία. Hello. Thank Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Η ακραία ανάληψη κινδύνου στον πιστοτικό τομέα και ιδιαίτερα στον, ε, σε τραπεζικές και επενδυτικές εταιρείες ε, έχουν συμβάλει στην χρεοκοπία και στην αποτυχία πολλών ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και το πρόβλημα αυτό βεβαίως έχει καλύψει, έχει εισβάλλει και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και πάρα πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η βασική επιτροπή για τα, τις κεφαλαϊκές απαιτήσει απαιτεί την αναθεώρηση όλων των προτάσεων και η Επιτροπή μας πρέπει να δώσει, να εκδώσει μια γνώμοδότηση η Επιτροπή μας, δηλαδή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Έχουμε λοιπόν υπόψη να κάνουμε μία επανεξιολόγηση των πολιτικών, των τραπεζών και των επενδυτικών εταιριών, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα το επεπτικό και ελεγκτικό σύστημα πρέπει να πω στην Επιτροπή, στην Κομισιόν δηλαδή, ότι ε, άρχισε πολύ καθυστερημένα το έργο της. Πολλές ζημίες και καταστροφές θα είχαν αποφευθεί αν είχαμε παρέμβει νωρίτερα. Τώρα αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι αυτή η καταστροφή δεν πρέπει να ξαναγίνει πιστεύω ότι ε, οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των προτάσεων της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Καταρχάς, λοιπόν, την καλύτερη διάθρωση των ε, αμοιβών, την καλύτερη μισθολογική διάθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ε, την επιβολή ενός, πιο, ενός βαθύτερου και πιο αυστηρού προφίλ διαφάνειας ε, που θα υποχρεώνει όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επενδυτικές εταιρείες ε, να προσφέρουν πρόσβαση ε, στα στοιχεία τους και στις πολιτικές τους. Επίσης, την καλύτερη διάταξη των αμοιβών και την υποστήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθολογικών πλαισίων. Ε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συστήσουμε ξεχωριστές μισθολογικές επιτροπές, επιτροπές που θα εξετάζουν ε, τα κίνητρα που δίδονται ε, στα διευθυντικά στελέχη και έναντι της ρευστότητα που υπάρχει στην εταιρεία θα πρέπει λοιπόν να δικαιολογήσουν μία εφικτή και βιώσιμη μισθολογική πολιτική. Επίσης, ε, θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση του, του ε, μετοχικού κεφαλαίου και την, ε, το, το, ότι θα πρέπει να λογοδοτούν τη λογοδοσία έναντι των επενδυτών και των κατόχων μετοχών, των μετόχων δηλαδή της εταιρεία. Και τέλος, ζητούμε να εφαρμοστεί μια ε, συγκριτική, ένα συγκριτικό πλαίσιο ελέγχου ε, το οποίο ε, προς το παρόν δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες οδηγίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά της εποπτείας και του ελέγχου που συνέβαλαν σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους διερμηνείς, λέει πολύ ευγενικά ο μιλητής, διότι μου είπαν ότι θα μπορούσα να μιλήσω ότι δεν θα μπορούσα να μιλήσω τη γλώσσα μου, δανέζικα δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη διερμηνία και γι' αυτό αναγκάστηκα να προετοιμάσω ε, την ομιλία μου, την παρέμβασή μου αυτή στα αγγλικά και δεί Και ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο για τους διερμηνείς, αλλά ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά τους και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Όντω υπήρχε πρόβλημα με την εξασφάλιση τη ιδανική δερμηνία και τελευταία στιγμή μόνο το μάθαμε, όπως και εσείς, ότι είχαμε τελικά δυσκολία με τα δανέζικα. Δυστυχώ, ήσασταν το υπόδειγμα και μιλήσατε τη γλώσσα του Σέξπιρ με άψογο τρόπο. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμά. Δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λεγιαρίκ για κοινή συζήτηση των δύο θεμάτων, 17 και 18, γιατί πρόκειται για δύο γνωμοδοτήσει. Βέβαια, μία θα δοθεί στην Οικονομική Επιτροπή και η άλλη στην Νομική Επιτροπή. Παρόλο που απευθύνονται σε δύο διαφορετικές επιτροπές, λοιπόν, τα δύο θέματα είναι συναφείω προς την ουσία του γι' αυτό και αποφασίσαμε να τα συζητήσουμε από κοινού. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Λεγιαρίκ για τα διοντολογικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των εταιριών. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολλές κυβερνήσεις ε, στον κόσμο και τα ίδια τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, καθώς και συνδικαλιστικά και κοινωνικά σωματεία, έκρουσαν το κόνδυνο του κινδύνου έναντι ενός νέου μηχανισμού που εμποδίζει τον, ε, τη λήψη απερίσκεπτου κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όπως διαπιστώνουμε εν μέσω της κρίσης και ενώ η ανεργία και η φτώχεια κλιμακώνονται, έχουμε και πάλι πληρωμή απερίσκεπτων και αστρονομικών πριμ ε, στα στελέχη. Και μερικές φορές τα πρίμα αυτα ξεπερνουν ξεπερούν κατά το βασικό μισθό ενός Γάλλου μισθωτού. Έχουμε και την περίπτωση των ε, χρυσών αλεξιπτώτων που συνεχίζονται να καταβάλλονται δαψιλώ. Όπως είπε ο κύριος Χρήστησεν στην αιτιολογική του έκθεση, το χειρότερο θα ήταν να αποφύγουμε την εφαρμογή κάποιων στοιχειωδών κανόνων εποπτικού και προληπτικού ελέγχου. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκύπτει στο θέμα αυτό, έστω και τώρα, και ασχολείται με τις διάφορες γνωμοδοτήσεις. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετήσω το δικό σας ρόλο και τη δική σας βούληση και αποφασιστικότητα να θέσετε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις στα τόσο επίκαιρα ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου του 2009 υιοθέτησε κάποιες συστάσεις για τα, τους μηχανισμούς αμοιβών και τις αρχές της διαφάνειας και διακυβέρνησης. Φυσικά αισθενιζόμαστε αυτές τις διοντολογικές αρχές, αλλά θα πρέπει πια να τις εφαρμόσουμε κιόλα. Συμφωνώ με τις διευκρινήσεις του κυρίου Κρίστενσεν ότι όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς θα πρέπει να υπάγονται σε αυτούς τους κανόνες και ε, να υπάρχουν υποχρεώμενες και κορυμμένες εξουσίες στις ελεκτικές αρχές. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια ζητήματα. Υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα εδώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε ένα οικονομικό μοντέλο που η αρχή της ανταγωνιστικότητας οδηγεί στην συνεχή αύξηση των αμοιβών των στελεχών που οι ίδιοι συνεχώς μειώνουν το μισθολογικό κόστος, το κόστος εργασίας, δηλαδή ε, περικόπτουν τους μισθούς και το επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Η αδικία και η ενισότητα είναι εμφανής και στην μεταβίβαση προς την ε, αποδοτικότητα του κεφαλαίου των μισθολογικών ροών. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων όπως λέω στο 2. Στο σημείο 3 ζητώ μια γνήσια διαφάνεια και για τις αποδοχές, καθώς και μια αναλογικότητα στην εξέλιξη αυτών των αμοιβών. Στα σημεία 7 και 9 επιμένουμε στην ανάγκη νέων δικαιωμάτων των εργαζομένων, των μισθωτών και των εκπροσώπων τους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για να εφαρμοστούν όλε αυτές οι αρχές και να λάβουν σάρκα και οστά και να μεταφραστούν και σε νομικό επίπεδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρηματοπιστωτικά κίνητρα, αλλά και κάποια νομικά εργαλεία με αυξημένο έλεγχο των εκλεγμένων οργανισμών, όπως ε, το, του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις Επιχειρήσεις, ε, του Συμβουλίου των Επιχειρήσεων. Άλλωστε, το Ελεκτικό Συνέδριο των Επιχειρήσεων έχει τη χάνει ε, κοινοτικής χρηματοδότησης. Επίσης, μπορούμε να προβλέψουμε ακόμη και ανάκτηση των με εφόσον αυτά καταβλήθηκαν για τη λήψη αποφάσεων που είχαν αρνητική επίπτωση είτε στο περιβάλλον είτε στην απασχόληση. Φυσικά το θέμα αυτό δεν εξαντλείται εδώ. Γι' αυτό και περιμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις και τροπολογίες σας για να τις συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λεγερικ. Η κυρία Καρή ζήτησε το λόγο. Διάβασα με προσοχή τα δύο σχέδια γνωμοδότησης και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω λίγο το ιστορικό. Λυπούμε που έφυγαν οι περισσότεροι συνάδελφοι, παρόλο που το θέμα αυτό ε, είναι κέριο. Το οικονομικό και, κλιμα... και οικονομικό κλίμα έχει επιδεινωθεί. Γίνονται μαζικές απολύσεις και μέσα σε δύο χρόνια αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση κόστησε σε 10 εκατομμύρια εργαζόμενους τη δουλειά τους, παρόλο που αυτοί δεν είχαν ζητήσει τίποτα. Και τι έκαναν οι χώρες, πηδαψίλευσαν κονδύλια στις τράπεζες και τα χρηματοστατικά ιδρύματα και έτσι οι πέτοι της κρίσης ε, έτυχαν κάποιες στήριξει. Το 2009 έπεσαν κατά 50% οι πιστώσεις. Ε, ε στο Παρίσι τα μπόνους φτάνουν στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ το 2008 είχαμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι απαράδεκτο γιατί ένας ε, ε, Γάλλος τρέιντερ θα πάρει 17 φορές 17 πλάσιο ε, επίδομα από ότι ένας μέσος Γάλλος εργαζόμενος. Δηλαδή όλα αυτά τα στελέχη λαμβάνουν πακτολούς χρημάτων ενώ οι εργαζόμενοι φυτοζωούν. Προτάθηκε από την κυρία Μέρκελ ε, να να φορολογούνται κατά 60% τα αστρονομικά μπόνους όταν ξεπέρνουν 25.000, αλλά δεν είναι αρκετές όλες αυτές οι προτάσεις. Δεν θα πρέπει να διονύσουμε τις ανεύθυνες συμπεριφορέ των φορέων του χρηματοπιστωτικού κόσμου που οδήγησε στην κρίση, την παρέτεινε και παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να ασχοληθούμε με το βασικό θέμα του καταμερισμού του πλούτου. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί που καταστρέφουν τον πλανήτη και περιβαλλοντικά δεν είναι οι πιο φτωχοί, αλλά οι πιο πλούσιοι, που είναι η βασική υπέτη για την επιδείνωση του κλίματος και του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, τα πρίμα παραμένουν σε αστρονομικά επίπεδα. Η διόρθωσή του είναι θέμα κοινωνική δικαιοσύνη και όχι μόνο περιβαλλοντική. Η κοινωνική κρίση δυστυχώ δεν έχει τελειώσει ακόμη, μάλλον τώρα αρχίζει και η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει το υπόδειγμα με τα μέτρα που θα λάβει. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κρίστενσεν για τη δική του γνωμοδότηση. Οι πράσινοι θα επιθυμούσε μεγαλύτερη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την πλαισίωση των, πολιτικών, των μισθολογικών πολιτικών. Και είμαστε υπέρ τη ολοσχερούς απαγόρευσης των χρυσών αλεξιπτώτων που δεν ανταποκρίνονται σε καμία οικονομική πραγματικότητα. Ζητούμε την σημαντική μείωση του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών κατά 20% επιπλέον της ετήσιας αμοιβή. Θα θέλαμε όλες οι καταβολές των μεταβλητών αμοιβών να γίνονται σε περιόδους και η καταβολή του πρώτου πριμ, του πρώτου μπόνους να μην γίνεται πριν τον πέμπτο χρόνο. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε την εξουσία των ε, μισθωτών σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των μισθολογικών ε, πολιτικών μια επιχείρηση και δίνοντα περισσότερες εξουσίες στις ε, επιτροπές του ομίλου και στις επιτροπές των εταιριών. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ξέφραγο αμπέλι για τους διοικητέ και τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων το θέμα και ούτε οι αποφάσει τους να διακυβεύουν τη βιωσιμότητα ολόκληρων επιχειρήσεων και να φέρουν σε δύσκολη θέση όχι μόνο τους μετόχους, αλλά και τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους επιχειρήσεις αυτές. Διάβασα με πολύ προσοχή και το εξαίρετο πόνημα του συναδέλφου Λεγιαρίκ και μάλιστα οι πράσινοι εστερνίζονται πλήρως ε, το περιεχόμενο της γνωμοδότησης και τις προτάσεις ε, του εισηγητού, του συντάκτου της γνωμοδότησης. Έχω δύο μικρές απορίες και προτάσεις. Η γνωμοδότηση μιλάει για θέματα δεοντολογικά σε σχέση με τη διαχείριση των εταιριών. Αυτό περιορίζεται μόνο στο θέμα των αμοιβών και των αποδοχών. Ε, είναι εσκεμμένος αυτός ο περιορισμός ή υπάρχει περιορισμός σε ό,τι αφορά το πεδίο, την εμβέλεια της γνωμοδότησης. Δεύτερη ερώτηση, για τις λοιπές αποδοχές. Θα ήθελα να είμαστε πιο ακριβείς στην τρίτη παράγραφο, σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο των μισθών στις επιχειρήσεις, καθορίζοντας ένα ενδεικτικό συντελεστή που θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, 40 φορές το μέσο εισόδημα στο ελόγο κράτος. Δεύτερη πρόταση να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή γνωμοδότηση και να συμπεριληφθούν τρία σημεία. Να επαναλάβουμε την προσήλωσή μα για την πάταξη οποιασδήποτε διακριτική μεταχείριση στη μισθολογική πολιτική και να προωθήσουμε την μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών, επιβάλλοντα κυρώσει στι επιχειρήσει που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση αυτή. Δεύτερη πρόταση, να υπενθυμίσουμε ότι η πάταξη των φορολογικών παραδείσων είναι προτεραιότητα και από την άποψη αυτή ο ρόλο των επιχειρήσεων θα είναι πρωταρχικό. Οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει δραστηριότητε ή επαφέ με μη συνεργάσιμα κράτη θα πρέπει να υπόκειται σε κυρώσει. Για παράδειγμα, να μην τη χάνει κρατικών ή κοινοτικών ενισχύσεων για μια τέτοια συμπεριφορά. Επίση, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλει μελέτη για τις ε, πρακτικές εξελίξεις σε θέματα δεοντολογίας στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και σωστό να ασχοληθούμε με αυτά τα κείμενα για λόγους τους οποίους έθιξαν ήδη και οι εισηγητές ιδιαίτερα όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσει οι οποίες μπορεί να βλάψουν και να ζημιώσουν μεγάλες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι οι παρατηρήσεις που έγιναν από τον συνάδελφο είναι πολύ σημαντικές και δεν είναι σύμπτωση ότι τον Απρίλιο του 2009 η Κομισιόν ήδη ανέφερε αυτό το θέμα, ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, δηλαδή ότι χρειάζεται ένα σύστημα ελέγχου, εποπτείας, το οποίο να ενισχύει και τη διαφάνεια. Όπως είπε και ο κύριος Κρίστενσεν, ε, εάν τα είχε πει αυτή η τα είχε όλα ε, πει η Κομισιόν νωρίτερα και τα έχει εφαρμόσει θα είχαμε ε, προλάβει ένα μεγάλο μέρος της καταστροφής. Πολλά ε, έχουν γίνει εντωμεταξύ βεβαίως διορθωτικά μέτρα, αλλά σε πολλά κράτη-μέλη το πρώτο που έπρεπε να γίνει είναι να αλλάξει νοοτροπία για να μπορέσουμε συνεχεία να λάβουμε θετικά μέτρα. Το συμπέρασμα είναι ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο και ίσως μπορούμε τώρα να προλάβουμε μελλοντικές ε, ζημιές, μελλοντικά σφάλματα, εάν προσαρμόσουμε και διορθώσουμε τα νομικά μας κείμενα και η πολιτική κατεύθυνση και βούληση στη χώρα μου προς αυτό κατευθύνεται, προς αυτή την προσέγγιση, δηλαδή ε, διόρθωση του νομικού πλαισίου. Μην ξεχνάμε όμως και την αντίσταση, διότι το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα είναι πάρα πολύ συντηρητικό. Είναι λοιπόν ε, απαραίτητο να επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Και επομένως και συλλογική αντιπροσώπευση και από αυτούς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και από αυτούς που εκπροσωπούν τους εργαζομένους. Και γιατί εμείς θεωρούμε δεδομένο κάτι που δεν είναι καθόλου δεδομένο. Δηλαδή, από τράπεζα σε τράπεζα, από πιστοτικό ίδρυμα σε πιστοτικό ίδρυμα, ε, διαφέρει ο τρόπος επικοινωνίας και Μάλιστα, μερικές φορές αυτή η διαφάνεια στην επικοινωνία αποτελεί ακριβώς στοιχείο του ανταγωνισμού. Ε, να σας πω επίσης ότι θα ήθελα να πω δύο πράγματα όσον αφορά αυτές τις, ε, αυτήν την τοποθέτηση Κρίστενσεν σχετικά με την έκθεση Καλά είναι όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορούν να εισαχθούν δεσμεύσεις όσον αφορά τις ποσότητες. Ε, γιατί η Moral Suasion νομίζω ότι λειτουργεί περισσότερο από την υποχρέωση και τη δέσμευση κυρίως ε, δε γιατί εδώ αντιμετωπίζουμε προσωπικές σχέσεις οι οποίες δεν πρέπει να ε, εκφυλιστούν και που από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούν να αναχθούν σε γενικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις γιατί αναπερίπτωση τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να ε, ενισχύσουμε την ε, ιδέα και τις ιδέες που ήδη εδώ αναφέρονται και προτείνονται. Δηλαδή, να υπάρχει ένα καλό σύστημα εποπτείας, το οποίο όμως θα συνοδεύεται και από ένα σύστημα κυρώσεων. μέσω τροποποιήσεων ε, ε, των οδηγιών όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο και όσον αφορά ε, την ιδιοκτησία. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για τα θέματα αυτά θα πρέπει να είμαστε και όταν μιλάμε για αμοιβέ ε, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ήδη είχε ξεκινήσει η συζήτηση αυτή από την Επιτροπή από τον Ζακ Ντελόρ. Το θέμα το οποίο είχε θέσει ο Ζακ Ντελόρ τότε δεν έχει λυθεί ακόμα. Συνέβη το εξή. Οι επιχειρήσεις για να έχουν ε, σύντομες ε, επιστροφές έκαναν, ε, δημιούργησαν ένα σύστημα το οποίο ε, απέδιδε σε πολύ βραχυπρόθεσμο ε, χρονικό, ε, σε πολύ βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα και επίσης ήταν ένα σύστημα το οποίο βασιζόταν στα μπόνους των στελεχών. Ήταν πραγματικά μια διαφορετική αντιμετώπιση της επένδυσης και επομένως μου αρέσει η αναφορά η οποία υπάρχει στο κείμενο του Λέζερικ η έννοια αυτή την οποία θέλω να ε, ενδυναμώσουμε περαιτέρω. Δηλαδή ότι η δυναμική απόδοσης θα πρέπει να αφορά όλο το, όλη την επένδυση και θα πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στην κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. γιατί διαφορετικά θα έχουμε συσταλτικές ερμηνείες διαφόρων ε, στοιχείων τα οποία θα αφορούν μονάχα αυτή την ανταπόδοση, ε, η οποία θα θεωρείται μάλλον ξεχωριστό κομμάτι από όλα τα υπόλοιπα. Ενώ η κοινωνική ευθύνη είναι καταμερισμένη και νομίζω ότι, μας, ότι δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας να γίνουν ταυτόχρονα οι δύο ε, συζητήσεις, να αντιμετωπίσουμε μαζί τα δύο θέματα αυτά. Επίσης, να αφήσουμε κάποιο χώρο στο χρονοδιάγραμμά μας, έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει στην αρμόδια επί Επιτροπή. Να δούμε τι γίνεται με την ε, γνωμοδότηση λέγαρικ. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλία τη Νομική Επιτροπή και μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι τα κείμενα τα οποία αναφέραμε ω κείμενα ε, αναφορά σχετικά με την απόδοση ε, και ε, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όσον αφορά τους μισθούς οπωσδήποτε θα αποτελέσει αντικείμενο της εργασία της Νομική Επιτροπής αλλά το εύρος της εργασίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί και επομένως ε, να μην τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα έτσι ώστε να περιορίσουμε τις δυνατότητες που θα είχαμε ενώ για την Επιτροπή μας ε, θα είναι μια πολύ πρώτη καλή ευκαιρία από την αρχή της θητείας ε, να συζητήσουμε θέματα διακυβέρνησης και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι τα ζητήματα αυτά και όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και όσον αφορά τη δυνατότητα απάντησης στην κρίση. Αυτό ισχύει και για την έκθεση του φίλου και συναδελφού Όλε Κρίστενσεν στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ε, ε, η κυρία Μακάρθη ασχολείται, συνεχίζει να ασχολείται με το θέμα αυτό. Δεν είμαστε δηλαδή μόνοι μας ε, και ούτε πρέπει να, είμαστε, να έχουμε φοβικά σύνδρομα. Θα πρέπει να μπορούμε να αναφέρουμε οτιδήποτε χρειάζεται να αναφέρουμε. όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση ε, Λεζιαρίκ, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. εάν ασχοληθούμε με δεοντολογία και όσον αφορά ε, και, και όταν ασχολούμαστε με, τις, με τους μισθούς και τις αποδόσεις ασχολούμαστε όχι για να δημιουργήσουμε κοινωνικά, κοινωνικούς αυτοματισμούς αλλά γιατί αυτού του είδους οι ε, μισθοί και αυτού του είδους οι αποδόσεις ε, ε, οθούν τα στελέχη σε ειδικέ συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις προς ζημίαν πλέον μακροπρόθεσμων και πιο μακρόθωρων πολιτικών και επενδύσεων. Εμείς δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο εναντίον των Golden Boys ή των Golden Girls. Νομίζω ότι η δημόσια συζήτηση εστιάστηκε υπερβολικά στα μπόνους. Το είπατε και στην γνωμοδότησή σας ε, όταν αναφερθήκατε στις συντάξεις. Ε, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα και να δούμε λίγο ε, την απόδοση μέσω καταμερισμού των stock options. Νομίζω ότι όλα αυτά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει επομένως να έχουμε μια πιο συνολική προσέγγιση της απόδοσης ή του μισθού. Επίσης, στον ε, τομέα αυτό, στον κλάδο αυτό, η συζήτηση γίνεται μεταξύ κωδικοποίησης, αυτορύθμισης, ε, νομικού πλαισίου κτλ. Εγώ νομίζω ότι ο ορισμός ενός πλαισίου ευρωπαϊκού ε, ευρωπαϊκού επίπεδου θα μπορέσει να μας ε, οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε εταιρεία, κάθε επιχείρηση στο όνομα της, ε, του ανταγωνισμού, στο όνομα της εθνικής νομοθεσίας ε, αρνείται, κρύβεται μάλλον πίσω από αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να αρνηθεί να ακούσει αυτά που λέμε εμείς. Οι ε, operators πρέπει να είναι σαφώς ορισμένοι από την Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ο καθορισμός ενός πλαισίου αναφοράς και ωφελήμων αρχών, ε, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό σημαίνει επίσης ότι από την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να σκεφτούμε μαζί τον τρόπο εποπτείας, πώς, δηλαδή πώς μπορούμε να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόζονται όλα αυτά σε κάθε κράτος μέλος. Και φυσικά όσον αφορά την ερμηνεία των συστάσεων από τα κράτη-μέλη και εδώ το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός όσον αφορά ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όσον αφορά τις χρηματιστηριακές ε, αγορές και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία. Αυτά και μέσω τροπολογιών βεβαίως ε, θα υποβάλω τις ε, σκέψεις μου. Έχω ακόμα ε, και άλλους αγορητές που έχουν εγγραφεί. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλτασάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Δύο λόγια θα πω. Είμαι και μέλος στην νομική επιτροπή, επομένως και εκεί με μεγάλη προσοχή θα ακούσω τι έχει να μας πει ο εισηγητής. Συμφωνώ απολύτως το πνεύμα και τη φιλοσοφία αυτής της γνωμοδότησης. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει κάποια ζητήματα να αποσαφινιστούν. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια γενική αναφορά στα νέα δικαιώματα των εργαζομένων που θα πρέπει να ταυτοποιηθούν στον, ε, στις σχέσεις ε, ανάμεσα ε, στις, εταιρείες, στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, ότι αυτή η σχέση ε, αφορά μονάχα την απόδοση, τη μισθολογική σχέση. Επίσης, θα πρέπει να δούμε καθαρά γιατί επιχειρήσεις μιλάμε. Μιλάμε για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μιλάμε για τράπεζες μόνο, μιλάμε για ε, εταιρείε τις οποίες είναι για επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο ή μιλάμε για καθαρά ιδιωτικές εταιρείε οι οποίες έχουν τελειώσει τελείως διαφορετικούς μηχανισμούς και τελείως ειδικό ε, τρόπο σκέψης και δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί σε αυτές να υπάρξει δυνατός ευρωπαϊκός έλεγχος. Το πεδίο εφαρμογής επίσης θα πρέπει να δούμε τι πεδίο εφαρμογής μπορεί να έχει αυτή η γνωμοδότηση, αυτή η θέση που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως θα πρέπει να κατανοήσουμε με ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους μπορούμε να ε, παρεύουμε με απλή θέση, με σύσταση σε, σε μια ε, οδό την οποία πραγματικά θα μπορούμε να ακολουθήσουμε και με μέτρα τα οποία πραγματικά θα μπορούμε από νομικής απόψεως εννοώ να πάρουμε. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ τελευταίος ο ομιλητής, πριν δώσω ξανά το λόγο ε, στον εισηγητή, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σωστό τώρα που όλοι έχουν φυγεί από την οικονομική κρίση να σκεφτούμε περισσότερο το θέμα της ε, επαγγελματική ηθικής στην οικονομία. Ε, ιδιαίτερα τώρα που ακούμε για αυτά τα τεράστια πριν των διευθυντικών στελεχών. Πρέπει όμως ε, να παραμείνουμε ρεαλιστές και να επιβάλλουμε μία ισόρροπη κατάσταση έτσι ώστε να μην ανταμείψουμε managers οι οποίοι έχουν ε, κάνει τεράστια σφάλματα στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα και πάρα πολλή αγανάκτηση στους πολίτες όταν βλέπουν να μείβονται αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τα τεράστια σφάλματα. Εμείς είμαστε συγγνωμοδότες, ε, δεν είμαστε η αρμόδια επιτροπή, αλλά ασφαλώς ακούγονται πολύ καλύτερες ε, προτάσεις από αυτές τις οποίες παρουσίασε η Κομισιόν όσον αφορά το προσωπικό και την ε, μισθοδοσία τους. Παραδείγματο χάρη ότι τα εργασιακά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λόγο στα πριμ και στα μπόνους των ε, managers. Πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως ε, λογικό διότι εκτός από τη διαφάνεια, τη διαφάνεια των μισθολογικών καταστάσεων, θα πρέπει να είναι σε θέση και εργασιακά συμβούλια και εργαζόμενοι να ελέγχουν ότι δεν θα ανταμυφθούν για τα σφάλματά τους οι υπεύθυνοι, αυτοί που τα έπραξαν και ότι τα πριν θα πάνε στους κατάλληλους ανθρώπους. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα υποβάλω μερικές ε, τροπολογίες και θα πρέπει πιστεύω να κάνουμε μια επανεξέταση της θέσης των, ε, της Επιτροπής αλλά προς την ίδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στους δύο συντάκτες γνωμοδότησης ε, με την ίδια σειρά που τους ακούσαμε και προηγουμένως. Πρώτα ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και ευχαριστώ όλες τις, όλα τα μέλη για τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλιά τους. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο αν και αυτή τη στιγμή, ακόμη και στην Ευρώπη, το πλαίσιο αυτό φαίνεται περιορισμένο. Ας πούμε ένα παγκόσμιο νομοθετικό πλαίσιο, μια, ένα παγκόσμιο πλέον κανονιστικό ε, πλαίσιο στο οποίο θα βασιστούμε για το μέλλον δεν έχω και πάρα πολύ εμπιστοσύνη στον τομέα αυτών, τον χρηματοπιστωτικό. Ε, αν δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή και αν δείτε και τις επενδυτικές εταιρείες, ε, νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχουν μάθει τίποτα. Ότι τα παθήματα δεν έγιναν διόλου μαθήματα. Ε, αν δείτε τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, αυτές οι τεράστιες ε, χρηματοπιστωτικές εταιρείε πληρώνουν αυτή τη στιγμή σήμερα μπόνους ε, των 500.000 δολαρίων τεράστια χρήματα λοιπόν στους ε, managers τους αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Βεβαίως ε, το επίπεδο των bonus δεν είναι, στο, είναι το ίδιο στην Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάσταση επικρατεί πάλι σήμερα. Έχει έχετε δίκαιο ότι ε, έχω ε, βασίσει ορισμένες ε, τροπολογίες μας στο έγγραφο της Κομισιόν, αλλά επίσης έχω απαντήσει και στο Συμβούλιο. Πολλά από, τα, από αυτά τα οποία έχω διατυπώσει βασίζονται στη θέση του Συμβουλίου. Ο κύριος Λεγιαρίκ. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι πολλές παρατηρήσεις από αυτές που ακούσαμε. Είχαμε σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη για τα θέματα αυτά. Και μάλιστα ακόμη και η G20 υπέβαλε στάσεις. Φαίνεται ότι απασχολεί αυτό το θέμα και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Και άρα, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, εμείς φέρουμε την ευθύνη ε, του προσδιορισμού ενός πλαισίου αναφοράς έως και ενός νομοθετικού πλαισίου αν γίνεται. Συμφωνώ με τις προσθήκες που πρότειναν συνάδελφοι. Τώρα για τη διαφάνεια. Υπάρχει δικαίωμα των μισθωτών που παράγουν αυτή την υπεραξία στις επιχειρήσεις να έχουν δικαίωμα επίβλεψης στις αποδοχές των στελεχών, των διευθυντικών στελεχών. Κύριε Μπαλτάσαρ, πρόκειται για δικαίωμα επίβλεψης στο σύνολο της διαχείρισης της επιχείρησης με τις ε, εδαφικές, ε, κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνέπειες που έχει διαχείριση αυτή. Τώρα το θέμα του καταμερισμού του πλούτου αρχίζει και αποκτά μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θετικό, θα πρέπει να εγκύψουμε στο θέμα του καταμερισμού του πλούτου μεταξύ των εργαζομένων των εισοδημάτων τους και των αποδοχών κάποιων διαθετικών στελεχών. Νομίζω ότι αυτό είναι μείζον θέμα και μας ενδιαφέρει και απόψη κοινωνικής και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Σε ό,τι αφορά το μεταβλητό σκέλος, αν συμφωνεί η Επιτροπή μας, εγώ είμαι υπέρμαχος της αυστηρής, του αυστηρού περιορισμού του μεταβλητού σκέλους. Και όπως είπε η φίλη Καρή Μαντελή, και εγώ προτιμώ να καθυστερήσει η καταβολή της συμπληρωματικής αμοιβή αποδοχής εφόσον αξιολογηθεί η προσφορά της. Επίσης, να μην ξεχνούμε και, το... και τη σχέση μεταξύ της αμοιβή των αποδοχών και της χρήσης των χρημάτων. Τι εξυπηρετούν τα κέρδη, την τροφοδοσία των φορολογικών παραδείσων, ενώ οι ίδιοι οι G20 είπαν ότι θέλουν να καταπολεμήσουν τους φορολογικούς παραδείσους. Προσοχή λοιπόν, τι χρηματοδοτεί το κέρδος. Συμφωνώ και στο σημείο αυτό με την κυρία Καρή Μαντελή. Θα πρέπει να φροντίσουμε, να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη τακτική έκθεση, ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση όλων αυτών των δράσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Διαδικαστικά τώρα, οι συντονιστές κατήρτσαν ένα χρονοδιάγραμμα και για τις διαγνωμοδοτήσεις ε, θα έχουμε προθεσμία τροπολογιών μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 12 το Μεσήλγι είναι ανταλλαγή απόψεων και τα δύο κείμενα θα εγκριθούν στις 16 και 17 Μαρτίου. Προτείνω να εγκρίνουμε καταρχήν το χρονοδιάγραμμα αυτό, αλλά θα το προσαρμόσουμε στη συνέχεια ανάλογα με τη... το ρυθμό μετάφρασης των ε, εκθέσεων κατ' ουσίαν. Γιατί αυτές, ε, αυτά τα κείμενα μας ενδιαφέρουν και πριν αποφαθούμε εμείς θα πρέπει να δούμε τις κύριες εκθέσεις πριν καταλήξουμε στις γνωμοδοτήσεις. Επίσης, θα πρέπει τις δικές μας γνωμοδοτήσεις να τις εγκρίνουμε πριν την ψηφοφορία της αρμόδιας κατ' ουσίαν επιτροπής. Αλλά πρέπει πρώτα να δούμε τα κείμενα. Πιστεύω ότι έτσι θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτή λοιπόν είναι καταρχήν η πρόταση για το χρονοδιάγραμμα. Διεκπαιρεώσαμε το πρωινό μας πρόγραμμα και σας δίνω ραντεβού στις 3